Colleagues, can I bring the meeting to all? Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε ποιον σας την ημερήσια διάταξη. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται για τις συνεδρίες των δύο επόμενων ημερών. Αν ναι, να προχωρήσουμε στην έγκριση των πρακτικών. Πρόκειται για τα πρακτικά της συνεδρίας της 18 και 19 Ιουνίου. Συμφωνείτε. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια Έχουμε την εφαρμογή της νομοθεσίας ε, του ενιαίου ουρανού. Η κυρία Φώστερ είναι η συγγήτρια. Ε, και οι δύο μαζί. Ένα, ένα, ένα, να το δούμε. Λοιπόν, καταρχήν να δούμε τον ενιαίο ουρανό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ όλους. Δεν θα μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες ε, για την επεξηγηματική δήλωση. Το έκανα αυτό την τελευταία φορά όταν ε, είχαμε τον πρώτο γύρο συζήτησης για τον ευρωπαϊκό ουρανό, αλλά να πω για τα μέλη που δεν ήταν παρόντα να εξηγήσω ότι η έκθεση αφορά την έκθεση της Κομισιόν για την νομοθεσία του ενιαίου ουρανού που λέγεται ε, «Καιρός να παρουσιάσουμε αποτελέσματα». Τι έκανα στην επεξηγηματική δήλωση και στο διατεκτικό ήταν να ενισχύσω τα μηνύματα ότι πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο και με μεγαλύτερη ταχύτητα σε ό,τι αφορά τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Έχουν ε, περάσει πάνω από 10 χρόνια από τότε που συμφωνήσαμε για τον κανονισμό σε αυτή την επιτροπή, όταν ήταν επίτροπος η κυρία Λογιόλαντο Παλάσιο και αποφασίσαμε ότι ήταν απαραίτητο να σκεφτούμε για το μέλλον. Ξέραμε ότι είχαμε κάποια προβλήματα τότε, μεγάλη συμφόρηση υπερβολική χορτικότητα κτλ. Και φυσικά μέσα στα 10 χρόνια σημειώθηκε πρόοδος. Έχουμε και την ε, κοινοπραξία του Σέζαρ. να δείτε την ανάπτυξη ορισμένων τιμάτων αυτού, έχουμε ε, και τον Τζόρτζα Ζεμπόφσκι, ο οποίος προσπαθεί ε, στα κράτη-μέλη να ασκήσει πίεση έτσι ώστε να υπάρξει κινητοποίηση σχετικά με το θέμα των λειτουργικών τμήματων του εναέριου χώρου. Και τέλος, αν ε, πρόκειται να έχουμε κάποιους πρακτικούς τρόπους προκειμένου να λειτουργούν οι επιχειρήσεις ε, και ο κλάδος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε εταιρείε που να έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχουμε την κατάλληλη χρήση του αέριου χώρου και θα πρέπει να έχουμε και τεχνολογία του 21ου αιώνα διαθέσιμη, έτσι ώστε όλοι να μπορούμε να αποφεληθούμε. Και τέλος, Πρόεδρε, νομίζω θα συμφωνήσετε ότι ο καταναλωτής ε, πληρώνει, πληρώνει εγκαίρος ε, και πληρώνει και το ύψος της τιμής. Τώρα έχουμε περιορισμένους πόρους, ε, αν δούμε τις ε, τιμές ε, του πετρελαίου και μπορούμε να κάνουμε το οτιδήποτε σε αυτό το κοινοβούλιο για να προωθήσουμε αυτά τα θέματα. Επομένως, πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και χάρηκα πάρα πολύ που ασχολήθηκα με αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση. Νομίζω ότι εξήγησα ότι εδώ μιλάμε για τη δημιουργία δεκάδων χιλιάδων θέσεων ε, εργασίας. Ε, μπορεί να έχουμε μεγάλη μείωση στις εκπομπές διεξοδίου του άνθρακα, γιατί φυσικά ε, αυτό θα είναι το αποτέλεσμα της πιο αποτελεσματικής χρήσης του ενέργειου χώρου και η ίδια η έκθεση χωρίζεται σε τρεις τομείς. Είχαμε την πολιτική συνεισφορά, είχαμε τη στρατηγική της ανάπτυξης και υπήρξε και ένα είδο συμπεράσματο ε, σχετικά με το τι πιστεύουμε ότι έπρεπε να κάνουμε. Είχαμε φυσικά και το χρονοδιάγραμμα που ήταν πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, να σας πω ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μάλα τους σκιώδεις εισηγητές. Τι κάναμε. Εγώ στην αρχική μου έκθεση προσπάθησα να διατηρήσω απλό το σώμα του κειμένου, να θα μπορούσα να έχω μπει σε πάρα πολλές λεπτομέρειες σε σχέση με το τι είναι το Σέζαρ και όλα τα υπόλοιπα, αλλά ουσιαστικά εδώ τι προσπαθώ να κάνω, να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στα κράτη-μέλη για να πούμε ότι τόσο καιρό πριν συμφωνήσατε για τον νέο ευρωπαϊκό ουρανό και τώρα πρέπει ε, να συνεισφέρετε με χρήματα και όχι με λόγια γιατί όλα αυτά καθυστερούν και πραγματικά για μας ε, ως βουλευτές ε, δεν είναι αποδεκτό να συμβαίνει κάτι τέτοιο αλλά ούτε και για τους συμπολίτες που ασχολούνται με αυτόν τον κλάδο. Έτσι λοιπόν, όπως σας είπα, ήταν ε, ειλικρινής και απλή η έκθεσή μου για το χρονοδιάγραμμα. Ρώτησα την Επιτροπή επί όλων των πτυχών και ζήτησα από την Επιτροπή να μας υποβάλει μια έκθεση τον Ιούνιο του 2012 γιατί θέλαμε μια επικαιροποίηση σε σχέση με το που βρίσκονται όλοι σε σχέση με την ανάπτυξη. Ξέρω ότι η κοινοπραξία του ΣΕΖΑΡ προχωρά συμμετέχει και ο κλάδος και όλοι συμμετέχουν και πρόκειται εδώ περί πολιτικής βούλησης. Αν δεν έχουμε πολιτική βούληση δεν έχουμε τίποτα. Πιστεύω ότι υπάρχει πολιτική βούληση. Τουλάχιστον η δική μου κυβέρνηση υποστηρίζει ένθερμα ε, αυτή την κοινοπραξία και είμαι σίγουρη ότι και οι συνάδελφοι από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη επίσης ασκούν πίεση στα δικά τους Υπουργεία έτσι ώστε όλοι να συμμετέχουν για να σημειωθεί κάποιο πρόοδος. Τώρα, Σχετικά με τις τροπολογίες, κατατέθηκαν αρκετές τροπολογίες. Νομίζω ότι οι περισσότερες ε, προσθέτουν αξία στην έκθεση. Καταλήξαμε σε αρκετού συμβιβασμού. Δεν νομίζω ότι πρέπει να σα του αναφέρω λεπτομερώ, ε, γιατί συζητήσαμε όλα αυτά τα θέματα μια μισή ώρα. Δεν υπάρχει λόγο να τα επαναλάβουμε εδώ. Έχουν συμπεριληφθεί οι απόψει ε, και του ΕΛΚΑ και των Σοσιαλιστών, των Πρασίνων, των Φιλελευθέρων και όλων και νομίζω ότι υπάρχει εδώ κατάληξη σε καταπληκτικούς συμβιβασμούς, σε καλούς συμβιβασμούς. Ε, κάποιες τροπολογίες όμως όπου μπορεί να μην ε, θα υποστήριζα την υπερψήφισή τους ε, αφορά κάποιε τροπολογίε όπου πιστεύω ότι ήδη οι πληροφορίε συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση. Δηλαδή δεν μπορούμε συνεχώ να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και θέλουμε να προσπαθήσουμε να έχουμε εδώ ένα συγκροτημένο κείμενο και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κανέναν, ούτε για τα κράτη-μέλη να πιστεύουν ότι υπάρχουν αμφισημίες. Δεν υπάρχει καμία αμφισημία, είναι ξεκάθαρα όλα τα μηνύματα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και τους σκιώδης εισηγητές που με υποστήριξαν τόσο πολύ και ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικοί σε σχέση με το να εκπονήσουμε μαζί τους συμβιβαστικές τροπολογίες. Και βέβαια πιστεύω ότι θα εξακολουθούν να υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι θα έχουν κάποιε ελαφρέ αποκλίνε απόψει, αλλά ελπίζω ότι αύριο στην ψηφορία θα έχουμε καλή υποστήριξη. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Φώστερ. Κυρία Ντεκού και το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα θα μιλήσω εκ μέρου του κύριου Μαρινέσκου, ο οποίο δεν μπορεί να παρευρεθεί εδώ διότι έχει σημαντικές υποχρεώσεις στη Ρουμανία, πολιτικές υποχρεώσεις. Θα είμαι σύντομος. Η ομάδα του ΕΛ και ο σκιώδης εισηγητής κύριος μαρινέσκου απευθύνεται στην κυρία Φώστερ. Πραγματικά σύνταξε μια πολύ περιστατωμένη έκθεση και η σκιώδης εισηγητής ε, ελήφθησαν υπόψη στις τροπολογίες. Πιστεύω πως είναι κοινό συμφέρον ο νέος ευρωπαϊκός ουρανός να θεσπιστεί τόσο όσο το γρηγορότερο δυνατόν και τα FABS, τα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου, είναι απολύτως απαραίτητα και πρέπει να τεθούν σε λειτουργία μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια, διότι όταν κάνουμε λόγο για την Ευρώπη και για αλλαγέ στην ε, δομή, τότε καταρχάς έχει να κάνει με την ε, εναρή ασφάλεια. Πρέπει να προσέξουμε τον τομέα αυτό και γι' αυτό είναι πάρα πολύ αναγκαίο να ε, τα λειτουργικά του μεταναέριου χώρου να υπάρχουν σε όλο τον ευρωπαϊκό ενέργειο χώρο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή ασφάλεια και σε περίπτωση ιδιωτικοποίηση να μην προκληθούν επιπλέον, ε, επιπλέον κόστος. Και είναι πολύ σημαντικό, όπως είπα, πρωτίστως ε, σημαντικό να ε, εγγυηθούμε την ασφάλεια στις απογειώσεις, στις προσγειώσεις, στις, στις μετακινήσεις στον ευρωπαϊκό Χώρο. Πρέπει να, το, να μπορούμε να το εγγυηθούμε αυτό και από τεχνικής πλευράς και από πλευράς προσωπικού, να υπάρχει πρόληψη ατυχημάτων. Αυτή είναι η κοινή μας ε, θέση και η κυρία Φώστερ ήδη το κατέστησε σαφές ότι πρέπει οι εθνικές μας κυβερνήσεις να χτίσουν μια γέφυρα όσον αφορά στις, ε, το στομέα των μεταφορών με το Υπουργείο Εσωτερικών τους και με τους ε, εθνικούς αρμόδιους Υπάρχει ανάγκη λοιπόν για, μια, για έναν συνολικό συντονισμό σε όλα τα στάδια και η μόνη λογική και συνετή λύση είναι πραγματικά αυτή που αναφέρεται εδώ. Διότι εάν δεν τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα πρέπει να δούμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν ανακοινώσει Όσον αφορά τα λειτουργικά τμήματα αέριου χώρου, τα FABS έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να συνεχίσουν εργάζοντας αυτά. Έχουν οριστεί εθνικοί εμπειρογνώμονες ε, και αναμένουμε την, την ε, έκθεση. Πρέπει όμως να παρατηρήσω δυστυχώς ότι δεν υπάρχει, δεν κινούνται πολύ τα πράγματα. Πρέπει να προβλεφθούν κυρώσεις για, όταν ε, τελούνται παραβιάσεις των συνθήκων. Το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε εμείς ως Κοινοβούλιο, ο κύριος Μαρινέσκου ως ισχύοντας εισηγητής πιστεύει ότι στην έκθεση αυτή αντιπροσωπεύεται καλά το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε και ότι υπάρχουν συμβιβαστικέ ε, τροπολογίες. Γενικά ο κ. Μανέσκου πιστεύει ότι καλύπτονται όλα τα σημεία, εκτός από ελάχιστα που χρήζουν ε, διευκρίνηση και πιστεύω ότι θα οδηγηθούμε σε καλή ψηφοφορία βασισμένη σε αυτά που έχουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Ντανέλη τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερως την συνάδελφο την κυρία Φώστερ και τους ε, συναδέλφους όδης εισηγητές για την ε, πολύ καλή έκθεση και την εξαιρετική συνεργασία που μας οδήγησε στο να πετύχουμε συμβαστικές τροπολογίες που στηρίζουμε όλοι. Ε, νομίζω έτσι καταφέρνουμε να στείλουμε με τον ε, καλύτερο τρόπο ένα ισχυρό μήνυμα προς την Κομισιόν, μία απέτηση να ασκήσει τις μέγιστες πιέσεις με άμεσες ενέργειες ώστε να επισπευθεί η εφαρμογή της νομοθεσίας του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού προς τα κράτη-μέλη. Ε, δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία οι προηγούμενοι ανέφεραν. Να πω μονάχα ότι μέσα από, την, ε, από τις συμβαστικές τροπολογίες ε, στηρίζουμε την αυστηρή στάση της Επιτροπής απέναντι σε όποια FABs δεν σεβαστούν την προθεσμία και όποια κράτη δεν προχωρήσουν σε αναγκαίες βελτιώσεις των σχεδίων επιδόσεών τους, ζητούμε την επίσπευση της στρατηγικής αλλά και της χρηματοδότησης για το ΣΥΖΑΡ και τέλος επισημαίνουμε τη σημασία του συστήματος επιδόσεων και φυσικά της στήριξής του. Κλείνοντας θέλω να πω ότι δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός σηματοδοτεί μια πραγματικά ριζοσπαστική μεταμόρφωση αέριας κυκλοφορίας Ευρώπης και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η προστιθέμενη αξία αυτής της, αυτού του σχεδίου, αυτής της νομοθεσίας μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου μέσα στο οποίο δεν υλοποιείται, δεν εφαρμόζεται αυτή η νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Mr. Thank you, I'm uh, Ευχαριστώ. Αντικαθιστώ τη συνάδελφο που ήταν σκιώδης σε αυτό το φάκελο και όπως ξέρετε το 2012 θα είναι σημαντικό έτος για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ουρανού <clears throat> και ε, η κυρία Φώστερ, ε, πιστεύουμε ότι έκανε μια πολύ καλή πρόταση και μπορούμε να υποστηρίξουμε και τις 21 συμβιβαστικέ τροπολογίες, αλλά και τις υπόλοιπες τροπολογίε. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι ε, ότι κατορθώνεται να, στείλνετε, να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα στα κράτη-μέλη, δηλαδή ότι τα ΦΑΜΠ ε, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο του 2012, αλλά θα πρέπει να έχουμε και κάποιες, ε, στο, κάποιους στόχους επιδόσεις που θα, επίδοσης που θα επιτευχθούν. Πολλά κράτη-μέλη παρουσίασαν κάποια εθνικά σχέδια επιδόσεων που δεν συνάδουν με τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως όμως ζητείται να αναλυφθεί δράση ε, για να επιληθούν αυτά τα προβλήματα και αν δεν σεβαστούν τα κράτη-μέλη την νομοθεσία ζητείται να ξεκινήσει η διαδικασία που παραβάσει. Επίσης ε, τώρα εργαζόμαστε επί ενός ε, πακέτου που συμπληρώνει αυτή τη δεσμή μέτρων και νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια πιο αποτελεσματική χρήση του ενέργου χώρου αλλά και των αεροδρομίων για να είναι ανταγωνιστική η Ευρωπαϊκή Αεροπλοία και για τις μολαντικές προκλήσεις. Ευχαριστώ κυρία και από τους Πράσινους. Ευχαριστώ πολύ. Έλαβα την ενημέρωση για όσα υπόθηκαν μέχρι τώρα. Θα συνεχίσω στα γερμανικά. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για όλες τις πληροφορίες. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα σημείο που θεωρώ πως είναι κεντρικό στα χρήματα. Τα χρήματα λοιπόν ε, απαιτείται σε αρκετές τροπολογίες ε, να διατεθούν ε, ευρωπαϊκά κονδύλια για τα FABs και για αρκετά πράγματα ακόμα. Τα ευρωπαϊκά χρήματα αυτή τη στιγμή δεν είναι πολλά. Και εάν δεν καταφέρουμε μέσα στις ε, συμβάσεις δημόσιου ιδιωτικού δικαίου να καταφέρουμε να, ε, δώσουμε, να συντάξουμε ένα δίκαιο μερίδιο, τότε το κόστος δεν θα καταναμηθεί δίκαια και ε, το κόστος θα το επομιστούν δυσανάλογα. Οι φορείς. Και πιστεύω πως αν γίνει αυτό δύσκολα θα οδηγηθούμε σε μια συμφωνία και έχουν γίνει τροπολογίες για αυτό, για ξεκάθαρους ξενώνες, για κανόνες, για δίκαιο καταμερισμό του κόστους, για fair share. Και διαφορετικά δεν μπορώ να φανταστώ δυνατόν να συμφωνήσουμε για τις τροπολογίες αυτές για όταν προβλέπονται να δοθούν περισσότερα ευρωπαϊκά χρήματα διότι η ιδιωτικοποίηση του κέρδους είναι κάτι που θεωρείται σύνηθες τον τελευταίο καιρό. Εδώ, ε, ο κλάδος των ενέργειων μεταφορών και ο νέος ουρανός ε, είναι αντικείμενο πολλών εθνικών συμφερόντων και πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε και να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα δεν θα ε, κατευθυνθούν προς λίγους συγκεκριμένους, αλλά με το fair share, με το δίκαιο κόστος. Τα εμπόδια στον ενιαίο ουρανό αυτή τη στιγμή έγινε στα κράτη-μέλη, στην ε, έλλειψη θέλησης ή στην έλλειψη δυνατοτήτων. Και πιστεύω ότι αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε βάζοντας το τσιρότο των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Δεν είναι λύση. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Σπρακ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συμφωνήσω ότι η έκθεση της κυρίας Φώστερ είναι πολύ καλή και πιστεύω να μπορέσουμε να βρούμε συμβιβασμό. Αυτός είναι ένας φάκελος ο οποίος έχει δείξει πόσο, πόσο εργατικό αποδείχθηκε το Κοινοβούλιο Βλέπουμε τα πλεονεκτήματα που έχει ο νέος ουρανός οικονομικά, αύξηση θέσεων εργασίας και συμφωνώ με την ε, εισηγήτρια ε, το να ασκηθεί πίεση στις εθνικές κυβερνήσεις για να γίνει πραγματικότητα ο νέος, εθνικός, ο νέος ουρανός. Ευχαριστώ για την Κομισιόν, κύριε Κασταλ, Κασταλέτη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να αρχίσω υπογραμμίζοντας για μία ακόμη φορά την ποιότητα της έκθεσης της κυρίας Φώστερ. Είναι εξαιρετική έκθεση, πολύ καλογραμμένη. τονίζοντας τα πραγματικά προβλήματα του Ενία ευρωπαϊκού ουρανού. Τώρα, όσον αφορά τι τροπολογίε που προτάθηκαν από ορισμένου από εσά, πιστεύω ότι στην πλειοψηφία του μπορούν να γίνουν αποδεκτέ από εμά. Καταλαβαίνουμε το σκεπτικό των τροπολογιών ότι στόχος του Single European Sky είναι η ασφάλεια και στις εταιρείε και στους επιβάτες, οι ποιοτικέ υπηρεσίες, οι πιο ασφαλείς υπηρεσίες, λιγότερο, ε, περισσότερο οικονομικές και υπηρεσίες οι οποίες θα οδηγήσουν στην ε, καλύτερη κατανομή του ενέργειου χώρου. Όσον αφορά τα FABs και, στην, και την ανάγκη να δημιουργηθούν όργανα διαχείρισης, αναγνωρίζουμε ότι είναι επίγουσα η εφαρμογή Η κρίση έχει οδηγήσει σε μία στάση της ανάπτυξης στον τομέα. Υπάρχει ανάγκη να εξυγχρονίσουμε το σύστημα και όσον αφορά τα FABs. Η Κομισιόν τώρα έχει στείλει υπενθυμίσεις στα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν τις απαιτήσεις, την ανάγκη μέχρι το Δεκέμβριο να έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις. Φυσικά η Κομισιόν προτίθεται να λάβει δράση προς τα κράτη-μέλη. Επίσης, αναθεώρηση των εθνικών σχεδίων. Ε, θα ήθελα να πω ότι τα εθνικά αυτά σχέδια υποβλήθηκαν πέρυσι τον Ιούνιο στην Κομισιόν και τότε η Κομισιόν εξέδωσε μία σύσταση σύμφωνα με την οποία τα κράτη-μέλη συνέταξαν ένα αναθεωρημένο σχέδιο. Τώρα η Κομισιόν στέλνει επιστολές στα κράτη-μέλη ζητώντας αυτά τα αναθεωρημένα εθνικά σχέδια. Τα σχέδια αυτά θα έλεγα πως οι γενικές γραμμές ε, ακολουθούν τους ε, στόχους που έχουν τεθεί. Χρειάζεται όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι ενώ ορισμένα κρατημέλη έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να φτάσουν σε αυτούς τους στόχους, ορισμένα άλλα κρατημέλη δεν το έχουν πράξει και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε στην επόμενη περίοδο αναφοράς που θα αρχίσει από το 2015 και μετά. Επίσης, focus την αύξηση της εγκατάστασης, στην ε, σύνδεση των ε, εθνικών υπηρεσιών, των πολιτικών, σύμφωνα με τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η χρήση του ΣΕΖΑ, ΣΕΖΑΡ θα ωφελήσει τις ε, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ορισμένοι από εσά ε, πρότειναν ομόλογα έργου για την χρηματοδότησή τους. Στον επόμενο γύρο οφείλουμε να διασφαλίσουμε την ε, επιμήκυνση του ΣΕΖΑΡ. Η έλλειψη πόρων και η ανεξαρτησία των ε, αρχών εξακολουθεί να είναι πρόβλημα. Ορισμένοι προτείνατε μία πιο κεντρική διαχείριση, όμως προτού γίνει αυτό πρέπει να αποσαφηνίσουμε τον ρόλο των κάθε, του κάθε Εθνικού Σώματος Διαχείρισης. Επίσης, η κοινωνική διάσταση και ο κοινωνικός διάλογος είναι σημεία κλειδί στην ανάπτυξη του τομέα. Επίσης, υπήρχε αναφορά στις ε, τροπολογίες για τη χωρητικότητα των αεροδρομίων. Φυσικά αυτές οι πρωτοβουλίες δεν αφορούν αυτή τη χωρητικότητα. Ξέρουμε ότι υπάρχει μία σύνδεση ανάμεσα στην εναέρια χωρητικότητα και στην χωρητικότητα των αεροδρομίων. Η χωρητικότητα των αεροδρομίων είναι κάτι που μπορεί να επηρεάσει την χωρητικότητα και την εναέρια κίνηση και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Θα ολοκληρώσω εδώ και θα ήθελα άλλη μια φορά να ευχαριστήσω την εξαιρετική δουλειά της εισηγήτριας και να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την έκθεση, το, η οποία μπορεί πραγματικά να δώσει όθηση στην εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Κομισιόν. θα είμαι σύντομη. Ξέχασα να αναφερθώ στη γνωμοδότηση της ΑΦΕΤ. Δεν θα σας δώσω λεπτομέρειες. Το, το περισσότερο κομμάτι το υποστηρίζουμε. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει μία παράγραφο την οποία δεν πρέπει να υποστηρίξουμε. Μου έκανε κατάπληξη διότι μιλάμε για τον ενιαίο ουρανό χρόνια και αποφάσισαν ότι χρειάζονται μία ε, αξιολόγηση επιδράσεων και αναρωτιόμουν γιατί δεν έγινε αυτό δέκα χρόνια πριν. Είναι βέβαια πολύ περίπλοκος ο, τομέας. Δεν πρόκειται όμως για διαστημικά θέματα. Λύνονται αυτά. Αλλά όταν αρχίζετε να διαβάζετε αυτή την παράγραφο, θα θα φανταζόσασταν ότι κάθε μαχητικό θα έπρεπε να εξοπλιστεί με κάτι διαφορετικά. Ε, μόνο τα μεταφορικά επιβατών χρειάζονται κάποιο εξοπλισμό βέβαια, ε, βεβαίως υπάρχει ένα κόστος, αλλά καταψήφισα αυτή την παράγραφο γιατί ήταν πολύ οπισθοδρομική και υπήρχαν αρκετές πληροφορίες στην υπόλοιπη γνωμοδότηση για να ξεχωρίσουμε τα επιβατικά από τα μαχητικά, τα πολεμικά δηλαδή. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Είχατε δίκιο που αναφερθήκατε στην χρηματοδότηση. Έχετε χρηματοδότηση από μία πλευρά και έχετε και τη χρηματοδότηση του Σέζαρ. Όλα αυτά είναι δημόσια, κρατικά έχετε βεβαίως θέματα έρευνας τεχνολογίας που εμπλέκονται. Δηλαδή δεν είναι ε, όλα τα λεφτά που προέρχονται από τον φορολογούμενο. Τίποτα δεν είναι δωρεάν βέβαια από την άλλη πλευρά, αλλά μακροπρόθεσμα πρέπει να πάρουμε τα ωφέλη και για τις επιχειρήσεις και για την βιομηχανία και για το καταναλωτή βεβαίως τελικά. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας Κομισιό. Ελπίζω να προχωρήσετε ε, με όλα τα πανιά ανοιχτά, ώστε να εξασφαλίσετε ότι όλα τα κράτη-μέλη ακούνε αυτό που λέμε. Έχετε όλοι μας την υποστήριξη προς αυτή την κατεύθυνση και ότι τυχόν ενέργειες λάβετε ε, για να ενισχύσετε το θέμα των FAB σας, παρακαλώ να τα αναλάβετε. Και θα περιμένουμε την έκθεση πρόοδου σας από σας αργότερα. Ευχαριστώ και ψηφίζουμε αύριο. Κυρία Φώστερ, όπως είπατε, λέει ο Πρόεδρος, αύριο ψηφίζουν στην, ψηφίζουμε στην έκθεση μεταφορών και στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πάλι κυρία Φώστερ, έχουμε να ασχοληθούμε με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Δορυφορικής Πλοήγησης. Ε, Τσάκη, έχεις το λόγο. Για να αλλάξω καπέλο. Λοιπόν, ε, θα ψηφίσουμε γι' αυτό που είναι καλή εκκίνηση. Θα ήθελα και πάλι λοιπόν, συνάδελφοι, να ευχαριστήσω την επικοδομητική στάση όλων. Μπορέσαμε να οδηγηθούμε σε ε, επικοδομητικές τροπολογίες συνεπώς. Υπάρχουν όμως και κάποιες τροπολογίες που δεν είναι του ίδιου τύπου. Θα ήθελα τώρα να επαναλάβουμε γιατί κοιτάμε αυτή την γνωμοδότηση. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε το GNSS να συνεχίσει. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε η χρηματοδότηση και όλα τα υπόλοιπα να υφίστανται. Δεν θέλουμε να έχουμε επικαλύψει. Θέλουμε τα δημόσια κονδύλια και είναι όλα αυτά δημόσια του φορολογούμενου να δαπανώνται σωστά. Και αυτό είναι ο ρόλο όλων των φορέων που ε, ασχολούνται με το GNS, ε, ο ρόλος που πρέπει να εφαρμόζουν. Τα ωφέλη του GNSS ε, βεβαίω είναι εντυπωσιακά και θέλουμε να συνεχίσουμε να τα έχουμε προφανώς και από τη δικιά μας την πλευρά τα ωφελήματα για το σύστημα μεταφορών τα οποία σας παρουσίασα στα σχόλιά μου όταν το πρώτο συζητήσαμε αυτό το θέμα, είτε πρόκειται για τις οδικές, συντηροδρομικές, συναυτιλια... Ε, θαλάσσιες μεταφορές. Όλα αυτά τα ωφέλη σημαίνουν ότι πρέπει να το σπρώξουμε να προχωρήσει. Χωρίς να μπω στις λεπτομέρειες υπήρξαν κάποιες παρανοήσεις. Ακόμη και εγώ χρειάστηκε να τα ξαναδώ, διότι όσον αφορά τα, ε, τη χρηματοδότηση είναι δημόσια, αλλά δεν είναι και τόσο σαφής διότι κάποιοι από εμά είμαστε εδώ και πηδάμε από ένα σχέδιο υποδομής σε ένα άλλο πρόγραμμα και μετά διαπιστώνεται ότι ορισμένε από τι τροπολογίες που έχουν υποβληθεί, που αναφέρονται στην χρηματοδότηση, κατά πάσα πιθανότητα αναφέρονται στον ορίζοντα του 2020 και πρέπει να διαφοροποιήσουμε ώστε οι τροπολογίες να έχουν πραγματικά σχέση με αυτή την έκθεση. Θα δείτε λοιπόν στον κατάλογο ψηφοφορίας ότι ενανύμαμε ε, αυτές τις πληροφορίες του συναδέλφους ώστε να μην θυγούν αν τυχόν δεν υποστηρίζουμε κάποια τροπολογία ακριβώς επειδή ε, η χρηματοδότηση δεν ήταν όπως την φαντάστηκαν. Ακόμη υπήρξαν θέματα όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες και τις περγολαβίες. Περγολαβίες λοιπόν. Αλλά και πάλι νομίζω ότι το ζήτημα είναι απλό. Δεν υπάρχει κανένας λόγο γιατί να μην υπάρχουν υπεργολαβίες αρκεί να εμπίπτουν αυτές τους σωστούς κανόνες, διεξαγωγής τους. Τελικά λοιπόν, θα έλεγα, ότι είχαμε μία λεπτομερή συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα πριν από μερικές εβδομάδες και γι' αυτό δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Δίνω το λόγο στους συναδέλφους. Ε, έχουν το σχέδιο ψηφοφοριών και ευχαρίστω ακούω τα σχόλιά τους. Πρόεδρος, ο κύριος Κάρον για το EPP. Ο κύριος Κούν, μάλλον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και την κυρία Φώστερ. Εξαιρετική η προετοιμασία των τροπολογιών, των 38 τροπολογιών έχουν ληφθεί υπόψη οι συμβιβαστικέ τροπολογίε οι γνωμοδοτήσει των Επιτροπών επί τη ουσία και πιστεύω ότι οι τροπολογίε μα έχουν συνταχθεί πολύ σωστά. Για μας το ΕΛΚ είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο συνάδελφο Μάρτιν Κίβετ είχε μια τροπολογία και έχει είχε εκφράσει κάποια σχολεία για την διατύπωση, αλλά του υποσχεθήκαμε ότι θα το προσέξουμε και θα συμπεριλάβουμε και το GNSS στην τροπολογία αυτή, ώστε να εφαρμοστεί στα αντίστοιχα άρθρα. Τροπολογία 44. Μετά, το κύριο σημείο το ανέφερε ήδη η κυρία Φώστερ. Πραγματικά, μέχρι σε, ποιο σημείο θα φτάσει η χρηματοδότηση συνολικά και αυτό είναι μια επένδυση. Είναι μια επένδυση από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατευθείαν στα κράτη-μέλη για, το σύστημα, για την δημιουργία του συστήματος Galileo. Έχουμε δώσει κονδύλια για το σκοπό αυτό και φυσικά είναι δικό μας συμφέρον να ξεκαθαρίσουμε ότι χρειαζόμαστε εφαρμογή του Γκαλιλαίου έτσι ώστε αυτή η επένδυση να αποδώσει εφαρμογή σε συγκεκριμένους τομείς, είτε στην ασφάλεια των, ε, των πλοίων, είτε για τα διόδια των ε, φορτηγών. Σε πολλούς τομείς μπορεί να εφαρμοστεί τον καλλιλέο. Υπάρχει μια ολόκληρη λίστα γι' αυτό. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμπεριληφθούμε στην έκθεση της Επιτροπής ΙΝΤΕ για την έξυπνη μεταφορά, για την αποφυγή της ε, κίνησης στα οδικά δίκτυα. Βέβαια, συνομιλήσαμε την Επιτροπή Ίτρα για τον προϋπολογισμό και συμφωνήσαμε ότι ότι οτιδήποτε που δεν εμπίπτει σε αυτές τις αμμοδιότητες θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Ευχαριστώ πολύ την ε, συνάδελφο. Θα λάβουμε την λίστα της ε, ψηφοφορίας και πιστεύω πως θα προχωρήσουμε καλά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Καλπεράρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και, τον, και την εισηγήτρια για τη δουλειά της ο Γιουροσλάβ δεν είναι εδώ, αλλά μου ζήτησε να πω δύο λόγια για αυτή την έκθεση. Γενικά μπορούμε να υποστηρίξουμε την νομοδότηση. Ο Μπόγκοσλαβ πάντως λυπάται ότι δεν έχει υπογραμμιστεί η ανάπτυξη των εφαρμογών που είναι το κρίσιμο στοιχείο για την φάση της εκμετάλλευσης. Δεν, ε, ε, δεν θεωρεί την ε, αφιέρωση κονδυλίων ε, δεν βλέπει μάλλον να αφιερώνονται κονδύλια για αυτή την ε, εφαρμογή ε, αναφέρονται περισσότερο κονδύλια μέσα στον ορίζοντα 2020 2020, αλλά όλα αυτά είναι πολύ ασαφή γιατί δεν ξέρουμε καν ποιο θα είναι ο προβολογισμός που θα αφαιρωθεί σε αυτόν τον ορίζοντα όσον αφορά την εφαρμογή. Για να σε σχέση με τα επιχειρήματα της κυρίας Φώστος, ο Μπογκοσλάβ Λιμπεράσκη υπέβαλε κάποιες τροπολογίες για να γίνουν τα πράγματα πιο εύκομπτα και για να μπορέσει η πρόταση αυτή να γίνει συμπληρωματική μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος για το 2020. Σας παρακαλώ λοιπόν να ρίξετε μια ματιά αν είναι δυνατόν σε αυτές τις τροπολογίες αλλά γενικά μπορούμε με τους συναδέλφους να υποστηρίξουμε τη γενική προσέγγιση. Και ο Ο κύριος Κλίντ ε, εξέταζε αυτή την έκθεση για μας. Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Συμφωνεί με την εισηγήτρια ότι ένα σύστημα δορυφορικής πλοήγησης θα μπορέσει να βοηθήσει και τους πολίτες και τις εταιρείες. Επίσης χαίρεται για την προσπάθεια ενίσχυσης της διαφάνειας όλες τις διαδικασίες και την ε, σωστή κατανομή ευθυνών και ε, ιδιαίτερα ε, τον ευχαριστεί το Κομισιόν θα αναφέρει στο Ευρωκοινοβούλιο. Πρέπει επίσης να γίνουν οι μεγαλύτερες προσπάθειες για την διαχείριση του προϋπολογισμού και του προγράμματος πιο αποτελεσματικά. Οι ιδιώτες επενδυτές δεν πρέπει να αποκλειστούν στην χρηματοδότηση αν το επιθυμούν. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Κυρία Κύριε Λίχτερμπεργκερ, ευχαριστώ. Σε γενικέ γραμμέ ε, με ικανοποιεί η έκθεση. Είμαι ικανοποιημένη και με, τις, με τους περισσότερους συμβιβασμούς. Ευχαριστώ όλους που ε, ανέφεραν την διαλειτουργικότητα και τον σημαντικό της ρόλο. Είχαμε μεγάλο έλλειμμα στον τομέα αυτό τα τελευταία χρόνια. Εάν είχαμε ασχοληθεί περισσότερο με την διαλειτουργικότητα, θα είχαμε γλιτώσει από πολύ σημαντικά προβλήματα ιδιαίτερα σημαντικό, θεμελιώδες μέρος. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω, όπως και πριν, το ζήτημα της χρηματοδότησης. Όταν δίνουμε χρήματα στις επιχειρήσεις, τους χαρίζουμε χρήματα, πρέπει να το λέμε με το όνομά τους και όχι να το κρύβουμε κάτω από τις ε, ωραίες διατυπώσεις, τη συγχρηματοδότηση η χρηματοδότηση είναι πολύ σωστή όταν τα project είναι καλά και ενδιαφέροντα. Όμως, σε αυτές τις ε, συνεργασίες πρέπει να κοιτάμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ για την Κομισιόν. Ο κύριος Νέιπηρ για την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την συγκεκριά για την εξαιρετική έκθεση. Νομίζω ότι είχαμε την τελευταία φορά ήδη την ευκαιρία να αναφέρουμε πόσο εκτιμούμε την έκθεση για τη σαφηνιά τη και επειδή προσφέρει υποστήριξη στο πρόγραμμα τα GNSS. Ακούγοντα ε, τι παρεμβάσει των βουλευτών σήμερα, βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο βαθμό ε, συνένεση. Υποστηρίζετε την πρόταση. Θα ήθελα όμω να αναφερθώ σε ένα στοιχείο που αναφέρθηκε από την κυρία Φώστερ και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα της χρηματοδότησης. Και θα τολμούσα να πω ότι κανείς μας εδώ δεν διαφωνεί με το πόσο αναγκαίο είναι να προωθήσουμε τις εφαρμογές. Και όπως ε, είπε κάποιος ευρωβουλευτής κάποια στιγμή, δεν έχει κανένα νόημα ε, η όλη υποδομή αν στη συνέχεια δεν υπάρχουν εφαρμογές. Όμως το θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι το πώς αυτές οι εφαρμογές τελικά θα χρηματοδοτηθούν και αν θα χρηματοδοτηθούν ε, με τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν δυνάμει αυτές τη νομοθετική πρόταση, ή αν θα αναζητήσουμε αλλού πηγές χρηματοδότησης. Ξέρετε ποια είναι η θέση μας σχετικά. Έχουμε υπολογίσει το κόστος, ε, τον προπολογισμό που παρουσιάσαμε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, μόνο για την εφαρμογή της υποδομής και κατόπιν οποιαδήποτε αφαίρεση αυτού για την ε, προώθηση ε, των εφαρμογών ουσιαστικά θα έθετε σε κίνδυνο την υλοποίηση ε, της υποδομής του Γαλιλαίου και του Έγκνος. Έτσι λοιπόν υπάρχουν και άλλοι λόγοι, αλλά τουλάχιστον για αυτό το λόγο αυτό υποστηρίζουμε απόλυτα την κυρία Φώστερ όταν προτείνει ότι η χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη και για τις εφαρμογές θα πρέπει να έρθει από το πρόγραμμα 2020. από το ορίζοντα 2020. Δεν θα χρονοτριβήσω. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω συνολικά για την υποστήριξή σας και ιδίω την κυρία Φώστερ για την εξωτερική έκθεση που εκπώνησε. Ευχαριστώ. Κυρία Φώστερ, θέλετε να επανέλθετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν κύριε επειδή αναφερθήκατε στις προφορικές τροπολογίες, ε, ήδη τις εξετάσαμε και τις έχουμε συμπεριλάβει στην, ε, στον κατάλογο της ψηφοφορίας ε, για να τις εξετάσουμε. Νομίζω ότι είναι ένας επικοδομητικός τρόπος να προχωρήσουμε, Πρόεδρε. Και τα σχόλια που ακούστηκαν από όλες τις ομάδες έχουν ληφθεί υπόψη για την αυριανή ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ. Αύριο είναι ψηφοφορία στην Επιτροπή και η Επιτροπή ΙΤΡΕ ε, θα ψηφίσει στις 6 Σεπτεμβρίου νομίζω και ελπίζουμε, είναι μόνο ενδεικτική ημερομηνία αυτή τη στιγμή, αλλά ελπίζουμε να ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Πολύ ωραία. Επόμενο σημείο στην Μερσή διάταξη αφορά το δέσμευμα μέτρων για τις χνοροθερίδες και εδώ έχουμε τον κύριο Ουγγίας ως εισηγητή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε σχέση με τον οδικό χάρτη που έχουμε καθορίσει, με το χάρτη πορείας, εγώ έχω προβλέψει να καταθέσω το σχέδιο της έκθεσης που διανεμήθηκε στους ε, Επιτρόπους και στους Σκιώδης και τους ευχαριστώ γιατί στα μέλη της Επιτροπής και στους Σκιώδης και τους ευχαριστώ για τη συνεργασία. Είχαμε και μια κρόαση όπου είχαμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις Θέλω να σας ρωτήσω πόσο χρόνο μου δίνετε πριν αρχίσετε να χτυπάτε το σφυράκι. Ξέρετε ότι διστάζω να λέω στους ηγητές ότι έχουν λίγο περισσότερο χρόνο από όσο έχει προγραμματιστεί, αλλά εντάξει. Εσείς ε, μπορείτε να έχετε λίγο χρόνο και αν ε, δω ότι μακρηγορείτε ιδιαίτερα θα προσπαθήσω και να σταματήσω. Αλλά αυτή τη στιγμή μας περσεύει κάποιος χρόνος. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Λέει ο Η έκθεση μου ουσιαστικά ακολουθεί τη λογική της παρέμβασης της Επιτροπής και συγκεκριμένα του Επιτρόπου Κάλλας και των υπηρεσιών του. για να είμαι συνθετικός. Υπάρχουν κάποιες κυρίες χαρακτηριστικές πτυχές. Καταρχήν, επειδή εισαγάγει τη δευτερογενή αγορά εμπορία των χρονοθυρίδων, ε, δηλαδή την εμπορία που όπως γνωρίζετε ε, σε ένα δεν ε, αναγνωρίζεται ως ε, νόμιμη σε όλα του Ηνωμένου Βασιλείου, αν και ως ένα βαθμό υλοποιείται. Έτσι λοιπόν ε, εισάγεται εδώ η νόμιμη αναγνώριση και με αντιστάθμιση μεταξύ, με αποζημίωση μεταξύ των εταιριών και αυτή η διαδικασία συνοδεύεται από κάποιες εγγύησεις, όπως παραδείγματο χάρη το χαρακτηριστικό της αμεροληψίας ε, του, της ρυθμιστικής αρχής, ε, του ρυθμιστή, ο οποίος ε, διορίζεται με έναν τρόπο έτσι ώστε να είναι αμερόληπτος απέναντι στις εταιρείε και απέναντι στις δομές των εδρομείων και απέναντι σε όλους τους συμμετέχοντες. Έτσι λοιπόν, εδώ έχει δυνατότητα να χρησιμοποιούνται κάποιες υπηρεσίες δρόμια σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σε μια συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Σε αυτό αναφερόμαστε όταν μιλάμε για σλότη, για χρονοθυρίδες. Εδώ έχουμε ουσιαστικά ένα τρόπο καθορισμού της φύσης ε, της χρονοθυρίδας, εισαγάγοντας μία έννοια που καθορίζει μία πλήρη, μία πολύπλοκη διάρθρωσή της. Και ουσιαστικά λέμε ότι αυτές οι χρονοθυρίδες θα δίνονται ε, για να εξυπηρετούν ε, τα συμφέροντα των πολιτών ε, που χρησιμοποιούν τις ε, αεροπορικές υπηρεσίες αλλά και που θα εξυπηρετούν και τα συμφέροντα των εταιριών αλλά και των αεροδρομίων. Καταρχήν πρέπει όμως να εγγυηθούμε να γίνει αντικείμενο σα πλήρης ανεξαρτησία του συντονιστή, του ρόλου του συντονιστή. Τι Τίθεται όμως ένα πρόβλημα ότι αυτός ο φάκελος όπως ε, συζητήσαμε την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε με τους Σκιώδης την περασμένη εβδομάδα, είναι ένας φάκελος ο οποίος παρουσιάζεται με ένα διαρθρωμένο τρόπο και εκεί παρουσιάζονται όλα τα προβλήματα της ε, ενέργειας κυκλοφορίας, προσφέροντας τη δυνατότητα ε, να αγγίξουμε όλες τις κύριες στοιχές από αυτή τη σκοπιά. Ένα θέμα που εξετάσαμε είναι το θέμα των σχέσεων μεταξύ των κόμβων και των περιφερειακών αεροδρομίων και των ε, περιφερειακών εδαφών γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτή τη σκοπιά ε, έχω καταθέσει μία πρόταση τροποποίησης στον κανονισμό που παρουσίασε η Κομισιόν που επιτρέπει τον ε, φορέα που χορηγεί τις χρονοθυρίδες να μπορεί να αρνηθεί μια εκχώρηση χρονοθυρίδας που θα ε, δημιουργήσει πρόβλημα στη σύνδεση ε, με τα περιφερειακά αεροδρόμια. Αυτό προϋποθέτει ότι κόμβει θα έχουν ε, τα κύρια αεροδρόμια δηλαδή, θα έχουν πάντοτε δυνατότητα να ευνοούν ε, τις διεροπηρωτικές συνδέσεις και να δημιουργούν ε, κάποιες συνθήκες ευνοϊκές για ε, την ε, σύνδεση με παραδοσιακές οδούς σύνδεσης, όπως το χάρη τη Βόρεια Αμερική και ε, με περιοχές αναδυόμενες όπως τις χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού. Και θέλω να κάνω δύο σκέψεις. Προβλέπετε ότι μέχρι το 2030 θα υπάρχει διπλασιασμός της ενεργείας κυκλοφορίας και ότι η χωρητικότητα των σημερινών χάπ, των σημερινών κόμβων δεν θα μπορεί να ικανοποιήσει τη ζήτηση. Έτσι λοιπόν για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς υπάρχει η επιτακτική απέτηση να αντιμετωπιστεί αυτή η αγορά, να ε, αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απαιτήσει. Θα είναι δύσκολο αυτό να γίνει με ε, μια πλέον άμεση λύση, δηλαδή με τον πολλαπλασιασμό ε, των hubs, των κόμβων, των νέων αεροδρομίων. Ε, εμείς ξέρουμε ότι είναι σχετικές οικονομικές δυνατότητες και το, το ότι ε, στην ε, Ευρώπη υπάρχει τέτοια κατανάλωση ε, δεν σημαίνει ότι θα επιφέρει και τις απαντήσεις. Έτσι λοιπόν εμείς προσπαθούμε να βρούμε τη βέλτιστη λύση. Δεν υπάρχει βέβαια κάποια λύση που να απαντά σε όλα, αλλά πρόκειται για μία πέντε, η οποία μας επιτρέπει στην περίοδο που αναφέραμε πριν να βελτιώσουμε το σύστημα το σημερινό σε ό,τι αφορά τη χωρητικότητα και θα μπορούσε να δημιουργήσει 60.000 νέες θέσεις εργασίας. Θα μπορούσε να γίνουν 60.000 νέες προ προσλήψεις και κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μία τελευταία σκέψη. Έχουμε αυτή την κατάσταση που σας περιέγραψα πριν και πρέπει να αποφασίσουμε αν πέραν από ε, τις αντιρρήσεις που εμείς ξέρουμε ότι υπάρχουν Υπάρχουν κάποιες αντιστάσεις, κυρίως από όσους ε, σήμερα ε, βολεύονται με την κατάσταση ως έχει από το status quo. Αναφέρουμε κυρίως σε κάποιες ε, αεροπορικές εταιρείες ε, που έχουν ουσιαστικά έρθει και έχουν αντικαταστήσει τις παλιές ε, εθνικές αεροπορικές εταιρείες. Αυτές επιθυμούν να μην αλλάξει τίποτα. Όμως κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα αρνητικό, θα ήταν καταστροφικό για την ενέργεια ευρωπαϊκή κυκλοφορία. Γιατί να παραμείνουμε τόσο ενεργοί ή να φανταστούμε λύσεις που δεν μπορούν να ελοπιθούν θα σήμαινε ότι καταδικάζουμε ε, τον ευρωπαϊκό χώρο ε, προς ε, την αποτυχία. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορούμε να επιτρέψουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ νομίζω ότι με την ε, συνεργασία που είχαμε και με τους Σκιώδης, ε, η οποία ήταν εξαιρετική, εξακολουθεί να παραμένει ανεκτός ο φάκελος και με την Κομισιόν έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια της προθεσμίας που έχουμε για την κατάσταση τροπολογιών, θα έχουμε τη δυνατότητα να διατυπώσουμε μια πολύ καλή πρόταση, να την υποβάλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, κ. Φλάντσα, για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν ε, να ευχαριστήσω τον συγητή για το έργο του μέχρι σήμερα. Όπως ξέρουμε, δεν είχαμε ένα έγγραφο εργασία για την έκθεση αυτή, όπως συνέβη για τους άλλους δύο φακέλους, για τα αεροδρόμια, αλλά είχαμε το κείμενο της έκθεσης, έτσι λοιπόν αυτό μας επιτρέπει να έχουμε πολύ συγκεκριμένες μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένε δυνατότητε κατάθεση τροπολογιών. Τώρα, να κάνω μια εισαγωγή. Βλέπουμε έναν κλάδο που, που συναντά πάρα πολύ μεγάλε δυσκολίε λόγω τη παγκόσμια ύφεση και όχι μόνο. Έχουμε κάποιες ε, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις παγκόσμιες αγορές ε, και προσπαθούν να αφαιρέσουν ε, από την Ευρώπη αυτό το κεντρικό χαρακτήρα του ενέργειου χώρου της και έχουμε μια κατάσταση ουσιαστικά κορεσμού. Και αυτό στα πλαίσια της ε, πρόβλεψης της αύξησης της ενέργειας κυκλοφορία τα επόμενα έτη. Έτσι λοιπόν πρέπει να φανταστούμε μία πολλαπλή απάντηση, μία απάντηση σε πολλά επίπεδα που δεν θα περιορίζεται σε μία δουλειά που πρέπει να κάνουμε μόνο για τα σλότ, αλλά και επί άλλων πτυχών. Εγώ νομίζω ότι ένα στόχο που θέτουμε είναι να αυξήσουμε τη χωρητικότητα του συστήματός μας, ώστε το στόχο αυτό θα πρέπει να το πετύχουμε με μια σειρά παρεμβάσεων και σκεφτούμε μία καλύτερη ρύθμιση για τις χρονοθυρίδες, αλλά επίσης σκέφτομαι και σημαντικές επενδύσεις ε, στις υποδομές, εκεί όπου φυσικά κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι συμβατό με την επικράτεια, με τα εδάφη και για το θέμα που συζητήσαμε πριν ε, σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του ενέου ουρανού και μια καλύτερη λειτουργία των FAB, των λειτουργικών τμήματων εναερίου χώρου γιατί κάτι τέτοιο θα διευκολύνει και τις ε, επιχειρήσεις ελέγχου του ενέργειου χώρου. Έτσι λοιπόν πρέπει να έχουμε μια πολλαπλή στρατηγική και οι χρονοθυρίδες είναι μόνο μία. Είναι μόνο ένα στοιχείο επί των οποίων πρέπει να εργαστούμε. Τώρα, σε σχέση με όσα βρίσκουμε ήδη στην έκθεση, το θέμα της αμεροληψίας της ανεξαρτησίας των συντονιστών μας βρίσκει σύμφωνους εμείς δεν έχουμε κανένα πιεστικό πρόβλημα σε καθημερινό επίπεδο με το ζήτημα αυτό. Ουσιαστικά δεν θεωρούσαμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά φυσικά υπάρχει το θέμα της ε, ανεξαρτησίας και της αυτονομίας της λήψης αποφάσεων και αυτό συνδέεται με το θέμα της χρηματοδότησης. Ποιος εγγυάται ε, το μισθό του συντονιστή. Ποιο πληρώνει το συντονιστή αυτό φυσικά είναι ένα θέμα και αν κατορθώσουμε να το αποσαφηνίσουμε και να προσδιορίσουμε πιο συγκεκριμένα ποιο πληρώνει τι και ποιον, τότε νομίζω ότι θα είναι πιο ανεξάρτητοι οι συντονιστές και θα βελτιωθεί το έργο τους. Συμφωνούμε λοιπόν για το θέμα αυτό, ό,τι αφορά τώρα τη δευτερογενή αγορά. Και εδώ Σίγουρα συμφωνούμε με την ανάγκη να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια. Θα πρέπει να πράξουμε έτσι ώστε η κατανομή των χρονοθερίδων ε, να μην δημιουργήσει μια αγορά αποκλειστικά οικονομικού χαρακτήρα, αλλά η ανταλλαγή των χρονοθερίδων είτε γίνεται με χρηματικό αντίτιμο είτε με παραχώρηση άλλων χρονοθερίδων να σημαίνει ότι θα έχουμε αύξηση της χωρητικότητας. Έτσι λοιπόν ε, να προσδιορίσουμε καλύτερα τα απαραίτητα κριτήρια της, διαφωνίας, ε, της διαφάνειας για να αναπτύξουμε το δευτερογενές εμπόριο νομίζω ότι είναι ένα χρήσιμο εγχείρημα. Σε ό,τι αφορά τώρα το νομικό ορισμό ε, της ε, χρονοθυρίδας, θα το συζητήσουμε αυτό και στο εσωτερικό της ομάδας μας. Εγώ συμφωνώ επί της αρχής, δηλαδή συμφωνώ με το να προσπαθήσουμε να ορίσουμε τι είναι το σλότ, αυτή η χρονοθυρίδα. Βέβαια προσωπικά ε, με προβληματίζει κάπως ε, η διατύπωση σχετικά με τον διατύπωση που έχει βρεθεί είναι η σωστή, γιατί θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιχειρησιακό επίπεδο σε στο να καταστήσει τα πράγματα πιο πολύπλοκα αντί να τα πλουστεύσει. Αλλά εγώ νομίζω ότι θα τα συζητήσουμε ξανά αυτά τα θέματα και στο ιστορικό της ομάδας μας, αλλά και με τους κοιόδης. Τώρα, κάτι που δεν υπάρχει ακόμη στην έκθεση. Εμείς έχουμε το μεγάλο θέμα της κατανομής ε, των χρονοθυρίδων, ε, το θέμα του κανόνα, χρησιμοποίησε τη χρονοθυρίδα ή θα την απολέσεις. Έτσι λοιπόν, αν ξεκινήσουμε από αυτή την αρχή, use it or lose it, εγώ συμμετείχα σε ε, όλες τις ακροάσεις ε, που ε, οργανώθηκαν από τον εισηγητή και από τις πολιτικές ομάδες, αλλά δεν κατόρθωσα να πιστώ για τους ορθούς λόγους της Επιτροπής. Εγώ νομίζω ότι αν βάλουμε στη ζυγαριά τις θετικές στοιχές που θεωρητικά θα μπορούσαν να προκύψουν από αυτή την τροποποίηση με με τις αρνητικές πτυχές που θα δημιουργούνταν από μια διαφορετική ρύθμιση σε σχέση με τους ε, υπόλοιπους πρωταγωνιστές σε παγκόσμιο επίπεδο, τελικά το πλεονέκτημα που θα ήταν η καλύτερη χρησιμοποίηση των χρονοθερίδων και αύξηση της χωρητικότητας δεν θα ήταν ε, τόσο υψηλό. Έτσι λοιπόν ε, έχω κάποιες αμφιβολίες σχετικά με το αν να τροποποιήσουμε αυτόν τον κανόνα σε ό,τι τώρα αφορά στο θέμα της ε, σειράς ε, των χρονοθυρίδων ε, έχω λιγότερο συντηρητική θέση. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε κάτι διαφορετικό, ίσως να συνδυάσουμε μία πρόβλεψη που να ισχύει με όλους με την δυνατότητα να χρησιμοποιούνται καλύτερα οι τοπικοί κανόνες, δηλαδή να έχουμε μία ελάχιστη πρόβλεψη για μία σειρά υποχρεωτική ε, σειρά χρονοθερίδων ε, που θα σέβονται όμως και τους τοπικούς κανόνες και θα επιτρέπουν στα τοπικά αεροδρόμια να διαχειρίζονται καλύτερα την ενέργεια κυκλοφορία. Επ' αυτού ευχαρίστως να το εξετάσουμε από κοινού. Και το τελευταίο ζήτημα σε ό,τι αφορά το slot reservation fee και τις κυρώσεις η Κομισιόν προβλέπει ένα τέτοιο τέλος που θα πληρώνουν οι ε, εταιρείε. Εγώ νομίζω ότι το να προσθέσουμε ένα επιπλέον κόστος ε, στις ε, αεροπορικές εταιρείες είναι κάτι επικίνδυνο, ενώ αντίθετα θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να εργαστούμε για να εγγυθούμε μια πραγματική χρησιμοποίηση του σλότ, δηλαδή να μην υπάρχει κατάχρηση της προ, ε, όταν προκλίνουν ε, την ε, χρονοθυρίδα και να χρησιμοποιείται σωστά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λέω κύριο ε, Σασόλη. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον συγγητή για το κείμενο που μας παρουσίασε. Ήδη σε προπροσκευαστικές συνεδριάσεις είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Όπως όλοι γνωρίζουμε πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, ευαίσθητο θέμα γιατί για τα αεροδρόμια, για τις αεροπορικές εταιρείε και για τους ταξιδιώτες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να διευκρινίσω αμέσω το εξή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το θέμα να υπάρχει ευρεία συμφωνία. Γιατί η δουλειά που θέλουμε να κάνουμε εμείς ε, είναι η εξής. Να κατορθώσουμε, να απελευθερώσουμε χωρητικότητα στα αεροδρόμια και να καταστήσουμε τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια πιο ανταγωνιστικά. Για το λόγο αυτό χρειάζεται ευρεία συμφωνία. Διάβασα με προσοχή την έκθεση και σε μεγάλο μέρος συμφωνώ. Θα ήθελα βέβαια να εμβαθύνω σε ορισμένε πτυχέ που κατά την άποψή μου θα έπρεπε να βελτιωθούν. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στη δευτερογενή αγορά εμπορία των χρονοθυρίδων, στον ε, ορισμό της χρονοθυρίδας ε, και στο ρόλο του συντονιστή. Ο όρος της ε, δημόσιας χρησιμότητας των χρονοθυρίδων. Θα έλεγα ότι εδώ θα πρέπει να είμαστε κάπως προσεκτικοί, γιατί θα μπορούσαν να προκύψουν παρεξηγήσεις. Παραδείγματο χάρη, για το ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να αποφασίσουν να διαχειρίζονται τις χρονοθυρίδες και να τις πολλούν όσο προσφέρει περισσότερα χρήματα και αυτό φυσικά θα προκαλούσε στρεβλώσει στην αγορά. Σε ό,τι αφορά τώρα στη δευτερογενή αγορά, να πω ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να κατανείμουν ένα μεγάλο τμήμα ε, των υποδομών και φυσικά αυτό συνδέεται και ε, με αυτό που είπαμε ε, για τη δευτερογενή αγορά ότι προκύπτουν από εκεί μεγάλα έσοδα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και με τις υποδομές για να ξεχρονίσουμε τα αεροδρομία, να δημιουργήσουμε νέα ε, χωρητικότητες, νέα χωρητικότητα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Θα πρέπει να είναι ουσιαστικά τα αεροδρόμια που θα διαχειρίζονται τα έσοδα προς αυτά. Αν δεν ε, προβούμε στη σωστή νομοθεσία, λοιπόν, στη σωστή νομοθεσία τότε ε, θα ε, αφήσουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να βάλουν αυτά τα χρήματα στον προπολογισμό και να μην χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για τη βελτίωση των υποδομών των αεροδρομίων. Σε ό,τι αφορά τώρα το ρόλο του συντονιστή. Νομίζω ότι εδώ θα έπρεπε να έχουμε κάποιε ρήτρε που θα εγγυώνται την ανεξαρτησία του συντονιστή και να ρυθμίζεται και πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Νομίζω ότι προ αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε, όπω κάναμε και σε μια προηγούμενη συνεδρίαση εισηγητή με τους κοιόδης εισηγητές να εργαζόμαστε και επί ε, του φορέα του Ευρωπαίου συντονιστή γιατί κάτι τέτοιο θα μας επέτρεπε να έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών μέγιστη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των χρονοθυρίδων στα κυρία αεροδρόμια της Ευρώπης. Αντίθετα, σε ό,τι αφορά τώρα τον κανόνα 80-20, νομίζω ότι όλοι συμφωνούν επί του εξή ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα τεχνικό ζήτημα. Σε ό,τι με αφορά, εγώ επιφυλάσσομαι, θέλω παραπάνω χρόνο για να κατανοήσω για το αν χρειάζεται ε, να, ε, να παρέμβουμε σε αυτό το θέμα γιατί στη συνέχεια τα προβλήματα θα αντικατοπτριστούν στους επιβάτες. Και, όπως είπε και ο συγητής, θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να αντιμετωπίσουμε τον κανόνα του 80-20 και τον αντίκτυπο που θα είχε αυτή η τροποποίηση στη σχέση μεταξύ της ευρωπαϊκής αγοράς με την παγκόσμια αγορά. Ίσως θα μπορούσαμε να οργανώσουμε το Σεπτέμβριο μια σειρά κροάσεων για να διευκρινίσουμε τα ζητήματα αυτά καλύτερα. Και κάτι τελευταίο, νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και ένα σύστημα κυρώσεων που θα είναι ορθά προσδιορισμένο για να αποθαρρύνουμε αθέμητες πρακτικές από την πλευρά των αεροπορικών εταιριών που θα αποφασίζουν να μην χρησιμοποιούν τις χρονοθυρίδες ή που καθυστερούν να τα επιστρέψουν, να τις επιστρέψουν τις χρονοθυρίδες. Πρόεδρε, Πιστεύω ότι η κατεύθυνση που ακολουθεί ο εισηγητής είναι σωστή. Με τη συνεργασία που προκλήθηκε μέχρι σήμερα από όλες τις πολιτικές ομάδες. Μάλιστα, ευχαριστώ κύριο Μπένιν για τους φιλελευθέρους. Yeah, I just, uh... uh ε, ήθελα βασικά να πω περισσότερα λόγια για μία παρατήρηση του κύριου Ουτζιάς. Να αναφέρθηκε στο θέμα των περιφερειακών αερολιμένων. Νομίζω ότι δεν μιλάμε μόνο για νησιά ή απομακρυσμένες περιοχές. Όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια απειλούνται αν ανοίξουμε την αγορά των χρονοτηρίδων υπερβολικά. Συνήθως υποστηρίζω λύσεις ανοιχτής αγοράς, ελεύθερης αγοράς για τα πάντα αλλά όταν υπάρχουν ελλείψεις στη λειτουργία της αγοράς, δεν το υποστηρίζω και εδώ μπορούμε να εντοπίσουμε ποια είναι η αδυναμία με την εξή έννοια. Από περιφερειακό σε περιφερειακό, με από κεντρικά αεροδρόμια σε κεντρικά αεροδρόμια έχετε αεροσκάφη με 300 και 400 επιβάτες. Από περιφερειακό σε περιφερειακό ε, ή από κεντρικό σε περιφερειακό 100-120 επιβάτες. Οπότε, αν θέλετε, η αρθριστική απόφαση μπορεί να μην είναι καλύτερη οικονομικά. Δηλαδή, τα αεροδρόμια, αν αφήσουμε την αγορά να λειτουργήσει ελεύθερα, μπορεί να εξασφαλίζει πολύ περισσότερες απτήσεις από κεντρικά σε κεντρικά αεροδρόμια και στη συνέχεια να αποκοπούν τελείως τα περιφερειακά αεροδρόμια από τα κεντρικά. Και όλα θα γίνουν αρνητικά δηλαδή. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν οριστικοποιήσουμε τη διατύπωση εδώ για την κατανομή των σλότ. Τα περιφερειακά αεροδρόμια πρέπει να έχουν πρόσβαση επαρκή στα κεντρικά Αλλιώς οι επιβάτες των περιφερειακών αποκόπτονται από τις πτήσεις μεγάλης διάρκειας, μεγάλων αποστάσεων. Πολύ ωραία να έχετε 300 πτήσεις μεταξύ Φραγκφούρτης και Λονδίνου με 300 επιβάτες ανά αεροσκάφος, αλλά αν δεν μπορείτε να φτάσετε στη Φραγκφούρτη, γενικά η ιδέα δεν είναι καλή. Θέλω να πω ότι εξατομικευμένες εμπορικές αποφάσεις για ένα σλότ χωρίς έλεγχο θα μπορούσε να σημάνουν την απαγόρευση τελικά των μικρών αεροσκαφών από τα περιφερειακά προς τα κεντρικά αεροδρόμια. Ευχαριστώ. Κύριος Λίχτενμπεργκερ. Η κυρία μάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, να αναφερθώ σε αυτό που ήδη υπόθηκε ανάμεσα στους συντονιστές των σχεδόν εισηγητών μιλάτε πάντα για ε, μεγάλους, ε, μεγάλα ποσοστά ανάπτυξης. Όμως η οικονομική κατάσταση και κυρίως η απώλεια εισοδήματος επηρεάζει επίσης και την αγορά εργασία για τους νέους. Τότε η ανάπτυξη, η, η, πώς, θα, πώς αναμένετε εσείς να τελεστεί η ανάπτυξη στους στους μικρούς αερομεταφορείς. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η ανάπτυξη χρειάζεται και προγραμματισμό και πολύ συγκεκριμένη στρατηγική για τους μικρούς αερομεταφορείς. Τώρα, όσον για τα περιφερειακά αεροδρόμια που ανάφερε ο συνάδελφος, πιστεύω, έχω την εντύπωση ότι μια αγορά η οποία τα τελευταία χρόνια είναι επακριβώς καταμερισμένη. Υπάρχει ένα μονοπόλιο, ένα ολιγοπόλιο στην Ευρώμη, Ευρώπη και εδώ οι περιφερειακές γραμμές κερδίζουν αρκετά χρήματα με την αύξηση των τιμών. Η κατανομή χρονοθυρίδων, από ό,τι μου λένε αρκετοί, είναι αρκετά επιλεκτική και είμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση όπου ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα μεγάλα αεροδρόμια είναι πολύ μεγαλύτερος, πολύ πιο έντονος και τα περιφερειακά αεροδρόμια δεν ε, βρίσκονται σε τόσο μειονεκτική θέση όπως λέει ο συνάδελφος. Όμως αυτή η αγορά που είναι τόσο επακριβώς ε, καταμοιρασμένη, η διαφάνεια και η ανεξαρτησία είναι οι δύο μεγαλύτερες ε, προϋποθέσεις, αν θέλετε, για μένα. Και όταν βλέπω πόσες πολλές προσπάθειες γίνονται για τη σύνδεση νέων αερομεταφορέων και, για την προ... και στις προσπάθειές τους να πάρουν μια θέση, αλλά δεν μπορούν να βρουν χρονοθυρίδες, τότε πρέπει να πω ότι τότε αυτό μου δημιουργεί υποψίες ότι πραγματικά υπάρχει μια έλλειψη διαφάνειας και ανεξαρτησίας. Και γι' αυτό η διαφάνεια και η ανεξαρτησία είναι οι δύο βασικότερες προϋποθέσεις που χρειάζεται να τεθούν από έναν συντονιστή. Για παράδειγμα, όταν έχουμε την ιδέα με, αυτήν την, το, το τέλος κράτησης ε, χρονοθυρίδας να δημιουργήσουμε έναν καλό μηχανισμό στην ε, αγορά. Εδώ πρέπει να βρούμε δυνατότητες να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα γίνει ε, αντικείμενο κατάχρησης από τους μεγάλους ε, μονοπωλιακούς αερομεταφορείς, αλλά θα υπάρξει η δυνατότητα και για νέες εταιρείες να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις χρονοθυρίδες και να περιορίσουν το μονοπόλιο να αποφευχθεί δηλαδή αυτή, αυτός ο θέμητος ανταγωνισμός ε, με τις τιμές. Όπως και στην δευτερογενή αγορά, έτσι και εδώ πρέπει να τεθούν κριτήρια για παράδειγμα, ο θόρυβο, τα επίπεδα του θορύβου, τα επίπεδα εκπομπών. Πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτά τα κριτήρια, διότι έτσι κι αλλιώ στι ενέργειε μεταφορέ, ακριβώ όπω και στι οδικέ μεταφορέ, η μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, ο στόχο τη μείωση είναι κάτι που αγνοείται, αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Διότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγνοείται παντελώς όσον αφορά το περιβάλλον. Και οι στρατηγικές που ακολουθούνται είναι ακριβώς αντίθετες. Γι' αυτό για μένα αυτή η ανταλλαγή, ναι, αλλά με κριτήρια, με προϋποθέσεις, έτσι ώστε τουλάχιστον, ε, όπως για παράδειγμα στον ενίο ευρωπαϊκό δεν υπάρχουν... Δεν, έχουν, δεν υπάρχει, έχει υπάρξει κάποια αλλαγή. Έτσι ώστε λοιπόν τουλάχιστον να υπάρχει κάπου μια μικρή ευκαιρία να ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Όμως, όπως είπα και προηγουμένως, για μένα το κεντρικό θέμα σε όλο αυτό το ερώτημα, σε όλη αυτή τη συζήτηση, είναι η διαφάνεια, η ανεξαρτησία, στην κατανομή των χρονοθερίδων, στον ορισμό των συντονιστών. Απόλυτα κεντρικό είναι αυτό, διότι η αγορά εδώ δεν λειτουργεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φώστερ. Τώρα. Ευχαριστώ, πολύ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή μας πραγματικά που οργάνωσε τα σεμινάρια, τις συναντήσεις των σκιωδών. Όλα αυτά καταδεικνύουν, καθώς και η συμμετοχή όλων των σκιωδών, καταδεικνύουν πόσο περίπλοκο είναι αυτό το θέμα. Μοιάζει ίσιο και απλό, αλλά δεν είναι. Σε όλες αυτές τις συζητήσεις λοιπόν οδηγηθήκαμε στις τοποθετήσεις των συζητήσεων που είχαμε πριν από χρόνια, παρόμοιες δηλαδή όταν ήμουν στο ΕΛΚ σε αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, ένας, ένα θέμα είναι ο νομικός ορισμός. Πρώτα απ' όλα δεν πιστεύω ότι είναι αυτός απαραίτητος. Δεύτερον, το σλότ είναι κάτι το αόρατο δεν είναι χειροπιαστό. Και αν θέλουμε να έχουμε δημοπράτηση, εμπορία, μπορούμε. Τώρα, γιατί αποφασίσαμε να το κοιτάξουμε αυτό και γιατί το κοιτάει και η Κομισιόν. Οπωσδήποτε είναι σημαντικό ο συντονιστής να μην μπερμποδίζεται. Και δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις. Είναι ανεξάρτητος. Και αν μιλήσετε με τους περισσότερους συντονιστές, πιστεύουν ότι έχουν την ελευθερία να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Και όταν δεν τους επιτρέπεται αυτό, οπωσδήποτε πρέπει να το διερευνήσουμε. Γενικά λοιπόν, συμφωνούμε όλοι με αυτό, δηλαδή αυτή την προσέγγιση για τον κανονισμό. Συμφωνώ με τον εισηγητή ε, και αναφέρομαι τώρα σε κάποιες λεπτομέρειες. Δεν πιστεύω όμως ότι χρειαζόμαστε ένα δίκτυο αεροδρομίων, δεν ξέρω τι υποτίθεται ότι αυτό θα είναι και συμφωνώ συνεπώς με τις σχετικές τροπολογίες. αφήσουμε τα πράγματα απλά. Επίσης δεν πιστεύω ότι πρέπει να είναι η διοκτησία των χρονοθυρίδων τα αεροδρόμια να έχουν την ιδιοκτησία των χρονοθυρίδων. Αυτό με φέρνει και στο ε, δευτερογενές εμπόριο. Όπως είπαμε στις συζητήσεις μας, ναι είναι δικιά μου χώρα και πράγματι στη δικιά μου χώρα έχουν δευτερογενή αγορά χρόνια τώρα. Ε, το 99% είναι ελεύθερο, το 1% είναι οικονομικό. Όσον αφορά τα κέρδη από αυτά, δεν νομίζω ότι θα πάνε ποτέ σε προγράμματα υποδομής, όλοι το ξέρουμε αυτό. Τα έσοδα θα... δεν ξέρω τι θα γίνει είναι εμπορική απόφαση, είναι εμπορικό απόρριτο και πρέπει κανείς να προσέξει πάρα πολύ αν το μεταβάλουμε, να μην οδηγηθούμε σε κάτι σκιερό όπου τα πράγματα δεν είναι διαφανή όπως είναι σήμερα. Βεβαίως εξαρτάται και από τη ρευστότητα της αγοράς για τις χρονοθυρίδες. Υπάρχουν δηλαδή πολλά τεχνικά ζητήματα τα οποία α, μοιάζει να είναι εύκολο να ρυθμιστούν αλλά δεν είναι και αυτονόητο. Αν, θέλουν τα κράτη, αν τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να υπάρχει δευτερογενής αγορά, να μην έχουν. Να είναι προαιρετική η απόφαση το 2020 παραμένει 2020. Νομίζω ότι λειτουργούμε μέσα σε ένα παγκόσμιο κόσμο, οι διεθνείς συμφωνίες και οι αποφάσεις λαμβάνονται για συγκεκριμένους λόγους. Δεν βλέπω, άμα κάτι δεν είναι σπασμένο, γιατί να το κολλήσουμε. Λοιπόν, το 2020 να μείνει όπως έχει και οι χρονοθυρίδες να μείνουν όπως λειτουργούν, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε τους τοπικούς κανόνες για κάποια αεροδρόμια. Όλοι οι πρωταγωνιστές συμφωνούν και ο συντονιστής παίζει ρόλο κλειδί. Τελευταία παρατήρηση, πρόεδρε. Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, θα θέλουν όλες οι διεθνείς εταιρείες να χρησιμοποιήσουν όλες τις χρονοθυρίδες τους για ε, υπερατλαντικές ε, πτήσεις. Βεβαίως θα θέλουν να τις χρησιμοποιήσουν, αλλά χρειάζονται και τους τροφοδότες. Δηλαδή χρειάζονται τα μικρά αεροσκάφη που θα φέρουν από τα περιφερειακά αεροδρόμια τους επιβάτες που θα πάνε στη συνέχεια στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα χρησιμοποιήσουν για διυπηρωτικές πτήσεις μόνο τις χρονοθυρίδες του, είναι λάθος μοντέλος, μοντέλο. Και βεβαίως πρέπει να προσέξουμε τις περιφερειακές περιοχές και πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Γενικά δηλαδή και πάλι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Και σίγουρα θα υποστηρίξουμε πολλές τροπολογίες που έχει υποβάλει ο εισηγητής. Ορισμένες δεν θα τις υποστηρίξουμε για τους λόγους που ανέφερα και σίγουρα θα λάβουμε υπόψη μας και τα υπόλοιπα σχόλια που θα γίνουν. Ευχαριστώ κύριε Σεγητά. Κύριο Ρίκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή ε, για το έργο του. Έχω μία ερώτηση. Δεν έχω απάντηση όμως. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση το γεγονός ότι σε σχέση με τις χρονοθυρίδες οργανώνουν μία πρωτογενή αγορά και μία δευτερογενή με κάτω από όρους που είναι τελείως αποσυνδεδεμένοι. Αυτό είναι μοναδικό διότι είτε μιλάμε για τα αυτοκίνητα δεύτερο χέρι ή για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υπάρχει μια διασύνδεση με τι πρωτογενούς και δευτερογενούς. Δηλαδή μπορεί να έχουμε ε, ε που να ορίζονται από τους συντονιστές στην πρωτογενή αγορά ε, κάτω από τους όρους οργάνωσης και ε, μύχιστοσποίησης, περιβαλλοντικούς κτλ. Δηλαδή εκεί έχουμε, αν θέλετε, προσδιορισμό βάση δημοσίου συμφέροντος και μετά περνάμε σε μια δευτερογενή αγορά που είναι τελείως ε, βασισμένη στο χρήμα. Έχω αμφιβολίες λοιπόν ότι σε αυτή τη δευτερογενή αγορά θα έχουμε μια ισορροπία που δεν θα είναι με βάση το χρήμα, δηλαδή θα, και εκεί θα έχουμε μεγιστοποίηση της κυκλοφορίας κτλ. Στη συνέχεια αναρωτιέμαι αν θα έχουμε πάντα ισόρροπες προσβάσεις, δηλαδή οι μεγάλες και σημαντικές εταιρείες θα μπορούν να επενδύσουν στη δευτερογενή αγορά διαστρεβλώνοντας την αγορά. Και ομολογώ, μου κάνει πολύ εντύπωση το γεγονός ότι θα οργανώσουμε μία πρωτογενή αγορά με έναν τρόπο και μία δευτερογενή με τελείως διαφορετικό τρόπο. Επίσης, και αυτή είναι ερώτηση προς την Κομισιό, όλη η αγορά θα γίνει δευτερογενής κάποια στιγμή, όπως αναφέρεται και αυτό κάπου στην έκθεση και μετά τι θα γίνει με την τρίτο γενή και τα λοιπά και μήπως σε δέκα χρόνια βρεθούμε σε ένα σύστημα το οποίο ε, δεν θα είναι καθόλου ευανάγνωστο οργανωτικά. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση η αταξία που εμφανίζεται στην οργάνωση των σλότς, πρέπει να σας πω στην έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, όπως ε, είχα πει και για το πακέτο αεροδρόμιο, αεροδρόμια, ε, έχω επιφυλάξεις και για την, τους κανόνες κατανομής των χρονοτηρίδων. Η βιομηχανία μας έχει δύσκολες αποφάσεις να λάβει, ιδιαίτερα ως προς τις θέσεις απασχόλησης. Αντιλαμβάνομαι την προσέγγιση της Κομισιόν, υπάρχουν θετικά στοιχεία, όπως η αναθεώρηση του νέου εισερχόμενου. Είμαι όμως επιφυλακτική ε, και το πάνε και άλλοι όσον αφορά την εισαγωγή δευτερογενούς αγοράς. Ασχολήθηκα λοιπόν με αυτό το θέμα πολύ προσεκτικά, διότι εδώ δεν πρόκειται να μπορέσουμε να μετρήσουμε απλά τα πράγματα και σκοτεινά. Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να θέσουμε για τη δευτερογενή αγορά είναι το εξής. Η δημιουργία της ανταποκρίνεται στο σκοπό τους, της χρονικής κατανομής για να αποσυμφορέσουμε τα αεροδρόμια μας. Δεν νομίζω ότι τα, η δευτερογενής αγορά δίνει την απάντηση. Πράγματι αυτή η μη μόνιμη νόμιμη αγορά υπάρχει σε κάποια αεροδράμια, αλλά δεν χρειάζεται να την νομιμοποιήσουμε. Δημιουργεί ανησυχίε. Μέσω πρόθεσμα, τι συμφέροντα έχουν οι εταιρείε να, να καλύπτουν περιφερειακές γραμμές που δεν αποδίδουν, ενώ θα μπορούν να πουλήσουν αυτά τις χρονοθυρίδες σε διεθνείς εταιρείες με υπερατλαντικές πτήσεις. Και οι τρίτες χώρες δεν θα έχουν τους ίδιους τους κανόνες αγοράς και θα έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό κατά των ευρωπαϊκών εταιριών όσον αφορά τις χρονοθυρίδες. Δεν βλέπω λοιπόν το συμφέρον για τη σύσταση μιας τέτοιας αγοράς. Ο στόχος μας είναι να έχουμε μία ανταγωνιστική αγορά με κανόνες ίδιους για όλους. Αυτή ε, για τη δευτερογενή αγορά κάποιοι είχαμε πει να φεθεί η ελευθερία στα κράτη-μέλη. Αλλά δεν μπορούμε από τη μία πλευρά να θέλουμε έναν νομισμένο ενιαίο ουρανό και μετά να διαφοροποιούμε τους κανόνες. Η άλλη πτυχή της πρότασης Κομισιόν συνεπάγεται την επιδείνωση των όρων χρήσης των χρονοθυρίδων. Μην ξεχνάμε ότι οι εταιρείε αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Και ε, ακριβώς αυτή τη στιγμή η Κομισιόν αντί να τις βοηθήσει ε, σκληραίνει τους κανόνες. Βεβαίως μπορούμε να βρούμε μια ισορροπία επιτρέποντας ε, μεταφορείς να αναπνεύσουν χρησιμοποιώντας καλύτερα και τις χρονοθυρίδες. Μου κάνει εντύπωση πως ο συνάδελφος Ουτζίας δεν τοποθετήθηκε πάνω σε αυτό. Ενώ οι τρεις προτάσεις λοιπόν της Κομισιόν πρέπει να γίνουν αντιληπτές και να τις διαπραγματοθούμε σαν ένα πακέτο αεροδρομίου, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις διατάξεις που εισάγουμε για το σύνολο της εναέριας κυκλοφορίας. Ε, αναφέρομαι στο ΕΤΕΣ για την αεροπλοεία, ε, μην επιβαρύνουμε τα πράγματα τόσο πολύ, να επιμικίνουμε την επέκταση των χρονοθυρίδων με επιβάλλοντας 95% χρήση συνεχή μου μοιάζει υπερβολικό. Πρέπει να βρούμε μια ισόρροπη κατάσταση που να αντανακλάται στην τελική έκθεση. Θα ήθελα ακόμη να πω ότι στην έκθεση του συναδέλφου Ιουζιάς βλέπω ότι προβλέπει μια κράτηση αυτών των χρονοθυρίδων ε, και θα πρέπει να ενισχύσουμε βεβαίως τις ποινές σε περίπτωση μη χρήση των κρατημένων χρονοθελίδων. Ε, ίσως η Κομισιόν θα μπορούσε να δημιουργήσει και ένα νέο επίπεδο με τα αεροδρόμια του δικτύου και όσον αφορά την αυτονομία του συντονιστή υποστηρίζω πλήρως αυτή τη θέση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι συνολικά όλοι συμφωνούμε, γενικά όλοι συμφωνούμε ε, ότι ε, θα υπάρξει αύξηση της ενέργειας κυκλοφορίας ε, και με τις κανονικές εταιρείε, αλλά και με τις εταιρείε χαμηλού κόστους. Θα πρέπει να βρούμε μια λύση προκειμένου να μην επιδεινωθεί αυτή η κατάσταση να μην επιδεινωθεί η κατάσταση τη ενεργειακής κυκλοφορία. Όμως νομίζω ότι εδώ θα τίθενται περισσότερα προβλήματα παρά παρουσιάζονται λύσει με διαφορετικέ αγορέ, όπω ε, είπε προλίγου, Κρικέ. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσδώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις προτάσεις που θα υποβάλουμε. Παραδείγματο χάρη, είναι αλήθεια ότι η θέσπιση των χρονοθυρίδων μου φαίνεται κάτι επικίνδυνο, όπως είπε και η κυρία Ντεβεράκη και άλλοι συνάδελφοι, και ιδίως αν λάβουμε υπόψη έναν ανταγωνισμό που θα μπορούσε να δημιουργηθεί μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιριών και των εταιριών που λαμβάνουν ε, επιδοτήσεις κυρίως από τρίτες χώρες. Θα πρέπει να προσέξουμε να μην καταστήσουμε πιο αδύναμο τον ε, ένα αέριο κλάδο μας, αλλά θα πρέπει να επιφέρουμε βελτιώσεις σε αυτή τη κυκλοφορία που θα είναι ένα και μεγαλύτερη και μας είπαν ότι και το 2030 αν δεν βρούμε την κατάλληλη λύση θα είναι τραγική η κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τώρα το να έχουμε αυστηρότερους όρους για τη χρήση των χρονοθυρίδων, οι νέες απαιτήσει ε, που προτείνονται μου φαίνονται κάπως ε, υπερβολικές. Ο κίνδυνος είναι να έχουμε εταιρείε που δεν θα σέβονται τα κριτήρια, δεν ε, θα θέλουν να εγκαταλείψουν τις χρονοθυρίδες τους ε, και θα υλοποιούν ε, πτήσεις με το αεροπλάνο άδειο Και αυτό θα έχει κόστος όχι μόνο για αυτή την εταιρεία, αλλά δεν θα είχε κανένα ενδιαφέρον ε, κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν ε, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με το να βελτιστοποιήσουμε τη χωρητικότητα των αεροδρομίων μας. Συμφωνώ με την ιδέα αυτή. Αυτό θα πρέπει να γίνει με συντονισμένη δράση και χωρίς να αποσταθροποιήσουμε τις εναερίες μεταφορές ε, που ήδη υφίσταται αρκετές ανατεραχές, ιδίως στους τελευταίους μήνες, τα τελευταία έτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Βλεστό. Ο κύριο Κράμερ. Για ε, Κύριε Ρικέ, αυτό ταιριάζει απόλυτα με αυτά που θέλω να πω. Μας είπατε γιατί χρειαζόμαστε δύο διαφορετικές αγορές. Στι συγκοινωνίε δεν έχουμε καμία αγορά απολύτω. Στην συγκοινωνία την θέσαμε την αγορά εκτό. Ό,τι χρειάζεται Ό,τι χρειαζόμαστε το επιδοτούμε, ό,τι μας είναι άχρηστο το φορολογούμε πάρα πολύ. Έτσι είναι τα πράγματα. Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια υπάρξει μια σημαντική αύξηση τη αεροπορική κίνηση. Και έχω πει πολλέ φορές 30 δισεκατομμύρια για τα καύσιμα κάθε χρόνο επιδότηση είναι πάρα πολύ. Οι αεροπορικές εταιρείε πρέπει να απαντήσουν στο εξή ερώτημα. Θέλουμε να ταξιδέψουμε, να κάνουμε τη δουλειά μας με λιγότερους επιβάτες αλλά με δίκαιες ε, τιμές ή με χαμηλές τιμές αλλά ψηλές επιδοτήσεις. Αυτό το πληρώνει και το περιβάλλον και ο φορολογούμενος. Γι' αυτό θέλουμε οικονομία της αγοράς. Όμως στην, ε, στις αεροπορικές μεταφορές είναι δυσανάλογο αυτό. Ένα φοιτητή, για παράδειγμα, που θέλει να πάει από το Βερολίνο στο τρένο, μου λέει ψάχνει στο ίντερνετ για την καλύτερη τιμή δεν τον ενδιαφέρει η εταιρεία. Και υπάρχει λοιπόν ω αποτέλεσμα μεγάλη πίεση στι χρονοθερίδε, υπάρχει μεγάλη πίεση στα αεροδρόμια, γι' αυτό θέλουμε την επέκταση. Αυτό μετά επιβαρύνει τη συνοδική κίνηση. Μετά από τόσα χρόνια, με τόσα δισεκατομμύρια ε, ε, επιδοτήσει, ακόμα έχουμε το πρόβλημα τη κίνηση. Και πιο μεγάλο από ό,τι πριν από 40-50 χρόνια. Γιατί λέγαμε τότε ότι ναι, οι οδικέ και οι οδικέ μεταφορέ πρέπει να αναπτυχθούν, χρειάζονται υποδομέ, τι λαμβάνουμε υπόψη. Όμω υπάρχουν παραδείγματα σε άλλα κράτη, σε άλλε πόλει, όπου η κίνηση έχει διαχειριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε έχει κερδίσει σε υποδομή και έχει μειωθεί. Πρέπει να προσέξουμε να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Φυσικά, θα πούν πολλοί ότι ναι, για παράδειγμα, θα σας πω ένα παράδειγμα. Πέταξα από τη Ρώμη στο Βερολίνο με 26 ευρώ, 25 και 99. Το λεωφορείο από τη Ρώμη στο αεροδρόμιο της Ρώμης κοστίζει 8 ευρώ. Το ταξί θα κόστιζε 50 ευρώ. Και καταλαβαίνετε πως αυτό είναι παρανοϊκό. Είναι όμως πραγματικότητα. Εάν θέλουμε να συνεχίσουμε, τότε κάθε 20 χρόνια πρέπει να αναθεωρούμε τα πράγματα. Και πρέπει να προσέξουμε, γιατί είδατε τι έγινε με, την, ε, με τη φούσκα των ακινήτων στην Ισπανία. Ό,τι, κατασκευα... Ό,τι είναι τεχνητό κατασκεύασμα κάποια στιγμή εκρήγνεται και αυτό κινδυνεύει να συμβεί και με, την, ε, και με τις εναέριες κυκλοφορίες. Και η κυβέρνηση που έχουμε τώρα στη Γερμανία, πριν από λίγο καιρό, ε, εισήγαγε ένα νόμο σχετικό με τις ε, δαπάνες της εναέριας κυκλοφορίας. 12 δισεκατομμύρια χρήματα φορολογούμενων ε, επενδύθηκαν. Έγιναν μετά περικοπές και όλες οι αεροπορικές ε, εταιρείες εξεγέρθηκαν στη Γερμανία. Και γιατί εξεγέρθηκαν, διότι έγιναν κατά ένα πολύ μικρό ποσοστό πιο δίκαιες αναγκάστηκαν να γίνουν πιο δίκαιες, να προσέξουν το περιβάλλον. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω ότι πρέπει να προσέξουμε, διότι αν συνεχίσουμε έτσι θέτουμε σε κίνδυνο το, μέλλον, το περιβάλλον, το μέλλον των παιδιών μας. Γι' αυτό πραγματικά στον εναέριο χώρο δεν χρειαζόμαστε πρώτογενή, δευτερογενή, τρίτο, τριτογενή ε, αγορά, αλλά έλεγχο και καθοδήγηση, αντικειμενικότητα και να δούμε πώς μπορούμε να κόψουμε την, ε, την κίνηση στο μισό και να έχουμε ε, ε, την ίδια και καλύτερη χωρητικότητα. Ο κύριος Λίντς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χίγγιν, συγγνώμη. Όταν άκουσα τους διαφορούς ομιλητές που μίλησαν ε, πιστεύω πως συμφωνώ με την Ζακλίν που μας είπε ότι ε, αυτό μας φάνηκε κάτι απλό στην αρχή. Όμως κάτι που φαίνεται απλό τελικά αποδείχθηκε πως δεν είναι απλό και ε, όσον αφορά το θέμα των ταχογράφων πιστεύαμε ότι ήταν κάτι τεχνικό και κάτι απλό, όμως ανακαλύψαμε πάρα πολλά διαφορετικά αντικρουόμενα, αντικρουόμενες λεπτομέρειες που οδήγησαν σε μεγάλες συζητήσεις ανάμεσα στα κρατημέλη και είδαμε ότι ήταν μεγάλο το θέμα. Yes, τέλος πάντων, πιστεύω ότι πρέπει να κοιτάξουμε την ουσία της έκθεσης και να τη δούμε, όπως είπε και η συνάδελφος Κριστίν και ο κύριος Βέστο, να δούμε ότι δεν έχει σκοπό η έκθεση αυτή να στραγγαλίσει την ανάπτυξη, αλλά να αυξήσει την διαφάνεια, να αυξήσει τον θεμητό ανταγωνισμό και την σωστή χρήση των ε, ισχυών των χρονοθερίδων. Και πιστεύω ότι ο εισηγητής της Κομισιόν έχει συντάξει ένα έγγραφο το οποίο αντικατοπτουρίζει αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε. Αν δούμε τις λεπτομέρειες, με την ε, πιθανότητα εισαγωγής της δευτερογενούς ε, αγοράς για τον ανταγωνισμό, να δούμε ότι ε, θα σα πω ένα παράδειγμα από το δική μου τη χώρα, από την Ryanair που χρησιμοποίησε αυτό το σύστημα. Εγώ δεν πετάω με τη Ryanair, αλλά η Ryanair με την πρακτική τη, ε, θέτει, ασκεί πίεση ε, στον εθνικό μα αερομεταφορέα, στην Lingus, στη Lufthansa και έχουμε δει ότι ο ανταγωνισμό έχει καλά αποτελέσματα. Είχε καλά αποτελέσματα σε αυτήν την περίπτωση. Ήταν προ όφελο των επιβατών. Έπειτα, η ενίσχυση της ε, διαφάνειας των διαδικασιών ε, απόδοσης χρονοθυρίδων. Φυσικά χρειαζόμαστε. Δεν την έχουμε προς το παρόν. Αυτό προτείνω να κάνουμε. Δεν βρίσκω κάτι λάθος. Μετά, η συμπερίληψη των ε, θηρίδων στο σύστημα αερίου ελέγχου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ουρανού. Πιστεύω πως είναι καλό και πως μας πάει μπροστά. Τώρα, Υποστηρίζω πλήρω ότι προς το παρόν έχουμε αραμέτοφορίς που κρατούν τις χρονοθυρίδες τους και στην τελευταία στιγμή λένε δεν τι θέλουμε και όταν κάποιο τότε θέλει να μπει στην αγορά έχει προβλήματα. Αυτό είναι αρνητικό για τον ανταγωνισμό. Αυτή η μη αποδοτική χρήση της υποδομής έχει οδηγήσει σε προβλήματα στην εισαγωγή νέων υπηρεσιών. Συμφωνώ με πολλούς από εσά για τις επιπτώσεις που θα έχει η πρακτική αυτή στα ε, μικρά, στα περιφερειακά αεροδρόμια, η ενίσχυση των κομβικών αεροδρομίων, διότι τα περιφερειακά αεροδρόμια είναι κλειδί για την επιβίωση των ίδιων των περιφερειών. και κινδυνεύουμε να έχουμε μεγάλο πρόβλημα στις περιφέρειες εάν δεν υποστηρίξουμε τα μικραπεριφερειακά αεροδρόμια. Όπως είπε και ο προηγούμενος συνομιλητής, εάν θέλουμε να έχουμε μια οικονομία της αγοράς, αυτό σημαίνει ανταγωνισμό και ο ανταγωνισμός είναι η ζωή του εμπορίου. Ευχαριστώ. Κύριε Μάισνερ, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, αυτό ο φάκελο με τις χρονοθυρίδε είναι το πιο περίπλοκο από όλο το πακέτο των αεροδρομίων. Μα φάνηκε στην αρχή απλό, εντάξει με το θόρυβο μπορούμε να δούμε τι θα κάνουμε, με με τις ονοθυρίδες αναρωτιόμασταν γιατί πρέπει να γίνεται λόγος γι' αυτό. Γι' αυτό όμως πραγματικά είναι ένα θέμα πάρα πολύ τεχνικό, πάρα πολύ περίπλοκο και που χρήζει εκτενού συζήτηση. Και όπως είπε ο συνάδελφος Κράμερ, φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς των αεροπορικών μεταφορών που επιδοτούνται. όντω, όμως δεν συμβαίνει μόνο εκεί. Και σε άλλους τομείς συμβαίνει αυτό και πιστεύω ότι ο κ. Σούτα έκανε πολύ καλή δουλειά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σκοπός μας είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας στα αεροδρόμια με τις προσγειώσεις στο 90, το 95% των χρονοδίδων στα αεροδρόμια είναι ήδη κλεισμένο. Επίσης πρέπει να δημιουργηθούν αίθουσες θέσεις εργασίας και στις αεροπορικές εταιρείες αλλά και στα αεροδρόμια. Δεύτερη άποψη. Μετά, ναι, μιλάμε σε γενικές γραμμές ότι αυξάνεται η ενέργεια κίνηση. Η ενέργεια Δυστυχώς δεν άκουσα αυτά που είπε ο κ. Κράμερ. Όμως πράγματι είμαι πεπισμένη ότι αυξάνεται και θα αυξάνεται η ενέργεια κυκλοφορία και πρέπει να αυξάνεται. Αλλά το ερώτημα του γιατί αυξάνεται κίνηση ενώ μειωνόμαστε ως πληθυσμό στην Ευρώπη, είναι πραγματικά κάτι το οποίο δεν μπορώ να εξηγήσω. Πρέπει να φροντίσουμε για το μέλλον των παιδιών μας και των παιδιών των παιδιών μας και τότε λοιπόν πρέπει να δούμε ε, και πρέπει να φροντίσουμε πώς θα έχουμε την καλύτερη δυνατή θέση. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε ιδιαίτερη προσοχή στις εναέριες μεταφορές και είδαμε με την πρόσφατη κρίση ότι ορισμένα Ορισμένοι κλάδοι προϊόντων, για παράδειγμα στη Γερμανία η BMW, δεν μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν όπως τώρα, διότι χρησιμοποιούν τις ενέργειες μεταφορές ε, για τις επιχειρήσεις τους και αυτό ε, είναι, κοστίζει πάρα πολύ. Στη Γερμανία η βιομηχανία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, όπως ξέρετε. Πέραν αυτού, πρέπει να μπορούμε να, κυκλοφο... να, κινούμε τα προϊόντα μας ελεύθερα, αλλά πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό χωρίς να αλλάξουμε ριζικά τα δεδομένα διαχείρισης. Και επίσης να αναλογιστούμε πώς εμείς με τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες μπορούμε να ανταγωνιστούμε τα, τις εταιρείες τρίτων κρατών που έχουν πολύ διαφορετικές ε, προδιαγραφές λειτουργίας και, πολύ διαφορετική, υπόκειται σε πολύ διαφορετική νομοθεσία. Για παράδειγμα, την Emirates. Είναι μια εταιρεία που ακολουθεί εντελώ διαφορετικές πρακτικές. Δεν μπορούμε εμείς να ακολουθήσουμε τις ίδιες πρακτικές, όμως πρέπει να την ανταγωνιστούμε. Και πρέπει λοιπόν να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στις χρονοθερίδες. Ποιος θα σε ποιον θα ανατίθενται οι χρονορθυρίδες, πώς θα ε, επηρεάσει, πώς δεν θα επηρεάσει αρνητικά την ε, εναέρια κίνηση. Ευχαριστώ κύριε Μάιστερ. Ο Μάικλ ξαναζητά το λόγο. Ένα λεπτό. Κάτι για τις θέσεις εργασίας. Από το 1994 στη Γερμανία οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά πολύ και κανείς δεν μίλησε γι' αυτό. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης χάθηκαν 70.000 θέσεις εργασίας και πρέπει να φροντίσουμε να επιβληθούν και κυρώσεις σε εκείνους που χρησιμοποιούν αθέμητες πρακτικές για τις θέσεις εργασίας. Πρωτού δώσω το λόγο στην Κομισιόν, θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια. Χάρηκα ε, που άκουσα ότι ο Μάικλ ε, Κράμερ γίνεται υποστηρικτής της οικονομίας της αγοράς. Ε, παρενέβη για να πω ότι η οργάνωση είναι πολύ διαφορετική μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς. Δεν είπα υπέρ ούτε κατά, ήταν λίγο αόριστο. Η κυρία Μέρα για την Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Ρικέ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους της Κομισιόν θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την σημαντική δουλειά που πραγματοποίησε και για το γεγονός ότι τόνισε την ανάγκη ανεξαρτησίας του συντονιστή χρονοθυρίδων. Επίσης υπογράμμισε και την ανάγκη για μια δευτερογενή αγορά για τις χρονοθυρίδες. Ευχαριστώ τον εισηγητή που δεν αμφισβήτησε την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη πειθαρχία εκ μέρους των αεροπορικών εταιριών στη χρήση της χωρητικότητας των αεροδρομίων. Βεβαίως και η ευελιξία είναι επιθυμητή, αλλά όταν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η χωρητικότητα έχει κορεστεί μόνιμα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή σε ώρες εχμής, τότε είναι πολύ σημαντικό συλλογικά να εξασφαλίσουμε οι αεροπορικές εταιρείε να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες τους βέλτιστα. Και η σειρά των, ε, η χρήση σειράς χρονοθυρίδων σε επίπεδο 95% και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 10 ε, το, χειμώνα, 15 το καλοκαίρι, αντί για 5 που προβλέπετε τώρα, ε, συνεχώς, ώστε να μην έχουμε καθυστερημένη επιστροφή των χρονοθυρίδων στο πουλ, στην ομάδα που είναι προς διάθεση, ε, πράγμα το οποίο συνεπάγεται ότι οι άλλες αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν πλέον. Λοιπόν, όλα αυτά ε, πρέπει να ακολουθούνται με κάποια συνέπεια. Όσον αφορά τώρα την δευτερογενή αγορά, αυτή πρέπει να ανταποκρίνεται στο δημόσιο συμφέρον. Επιτρέψουμε στις αεροπορικές εταιρείε να πολλούν και να αγοράζουν χρονοθυρίδες, θέλουμε να το πράξουμε για να αφήσουν να ελευθερώσουν χρονοθυρίδες οι οποίες να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν από άλλες εταιρείε που ενδεχομένως θα τις χρησιμοποιήσουν καλύτερα. Δηλαδή να μπορέσουν να πάνε προς τη ζήτηση οι χρονοθυρίδες, τη ζήτηση που όπως την εκφράζουν οι επιβάτες. Οι μελέτες που ζητήσαμε καταδεικνύουν ότι οι δευτερογενείς αγορά των χρονοθυρίδων επιτρέπουν σε περισσότερους επιβάτες να ταξιδέψουν μέσα στη χρονιά. Δηλαδή, συν 14 εκατομμύρια επιβάτες έχουμε το χρόνο, χάρη στην εισαγωγή της δευτερογενούς αγοράς χρονοθυρίδων στην Ευρώπη. Θα είχαμε, αν το πράξουμε. Ήθελα επίσης να επισύρω την προσοχή σας ότι ορισμένες τροπολογίες όπως είναι διατυπωμένες αυτή τη στιγμή μπορούν να υπονομεύσουν την αποτελεσματικότητα αυτού του μηχανισμού της δευτερογενούς αγοράς. Πρώτα απ' όλα δίνοντας ένα κομμάτι των εσόδων στα αεροδρόμια. Αυτό αποτρέπει τις αεροπορικές εταιρείες από την πώληση των χρονοτηρίδων. Εμείς θέλουμε να μπορέσουν να πουλούν και να αγοράζουν οι αεροπορικές εταιρείες. Εισάγοντας λοιπόν μία υποχρέωση απόδοσης των εσόδων στα αεροδρόμια, μπορούμε να μπορεί να υπονομεύσουμε το σύστημα. Να μην λειτουργεί σωστά δηλαδή. Το ίδιο ισχύει και με τις οικονομικές ροές που πρέπει να είναι πιο διαφανείς. Συμφωνούμε απόλυτα με αυτό που λέει ο εισηγητής, να ενισχύσουμε τη διαφάνεια όσον αφορά τις ενέργειες του συντονιστή. Πιστεύουμε όμως οι ατομικές συναλλαγές μεταξύ αεροπορικών εταιριών δεν πρέπει να δημοσιεύονται. Το συνολικό αποτέλεσμα ναι, για την ενημέρωση όλων. Αλλά οι συγκεκριμένες συναλλαγές δεν χρειάζεται να δημοσιοποιούνται, θα μπορούσε αυτό να δημιουργήσει πρόβλημα. Μία τροπολογία αναφέρεται στη συνδεσιμότητα και την πρόσβαση στα αεροδρόμια που δεν είναι συντονισμένα. Και έρχομαι τώρα στο θέμα του περιφερειακού και την εξυπηρέτηση των περιφερειακών αεροδρομίων που είναι πολύ σημαντικό ζήτημα όταν μιλάμε για δευτερογενές εμπόριο ε, των χρονοθυρίδων. Λοιπόν, το δευτερογενές εμπόριο μπορεί να οδηγήσει στο άνοιγμα νέων ε, δρομολογίων μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας το υπενθυμίζω αυτό. Υπάρχει αυτή τη στιγμή εταιρείε που θέλουν να εξυπηρετήσουν κάποια δρομολόγια, αλλά επειδή όμως δεν υπάρχει κινητικότητα στα σλότ, υπάρχει πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, δεν αμφισβητούμε ένα σύστημα το οποίο λειτουργήσε καλά. Η υποχρέωση δηλαδή δημόσιας υπηρεσίας. Το σύστημα όπως έχει διατυπωθεί μέσα στο πλαίσιο της πρότασής μας και του κανονισμού που εισάγει ε, την εσωτερική αγορά αεροπορικών μεταφορών του 2008 ε, μπορούμε να προσφύγουμε στο δημόσιο συμφέρον πάντα. Λοιπόν, έχουμε για να εξυπηρετήσουμε τις ενδοκινοτικές ε, γραμμές έχουμε ενισχύσει την έννοια του νέου εισερχόμενου. Ο εισερχόμενο είναι μια εταιρεία που έχει τέσσερις τέσσερα δρομολόγια την ημέρα προς πίσω, 9 χρονοθυρίδες και μπορεί να επωφεληθεί από την κατανομή της ομάδας προς κατανομή. Και στο επίπεδο του χαρτοφαλοκίου του νεοεισερχόμενου μπορεί να αυξήσει 5 με 10%. Δηλαδή, με άλλα λόγια, στην πρότασή μας θελήσαμε να εξασφαλίσουμε τις βέλτιστες δυνατόν συνθήκες για την περιφερειακή εξυπηρέτηση, θεσπίζοντας μηχανισμούς αγοράς για να παρακολουθήσουμε τη ζήτηση. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκαν πολλοί βουλευτές. Ειδικότερα το θέμα των αεροπορικών εταιριών τρίτων χωρών και του κινδύνου ορισμένες εταιρείες που ενισχύονται, επιχορηγούνται να αγοράσουν πιο εύκολα χρονοθυρίδες από κοινοτικά αεροδρόμια, ενώ οι δικές μας αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν μια δυσχερή οικονομική κατάσταση. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τις σχέσεις μέσα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τις αεροπορικές υπηρεσίες. Αυτή είναι και η ουσία του θέματος. Δηλαδή, όταν ένα κράτος μέλος διαπραγματεύεται δικαιώματα κυκλοφορίες, διαπραγματεύεται και κάτω από άλλες, άλλους όρους. Και το ίδιο κάνει και η Κομισιόν όταν διαπραγματεύεται για εναέριες υπηρεσίες. Συνεπώς αυτή η υπόθεση έχει σχέση με τη διαπραγμάτευση αυτή και όχι με τις χρονοθύριδες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να δώσουμε το λόγο και πάλι στον κύριο Σιγητή για τα συμπλασματικά σχόλια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι τα σημεία που αναφέρθηκαν από τους και και από τους συναδέλφους που πήραν το λόγο έδωσαν, ε, σας έδωσαν μια ιδέα για το πόσο πολύπλοκο είναι το ζήτημα. Ουσιαστικά με το ρολόι στο χέρι δεν ε, ε, πρόκειται να δώσουμε συγκεκριμένα λεπτά για την απογείωση και την προσγείωση σε έναν αεροδιάδρομο. Δεν πρόκειται περί αυτού, αλλά μιλάμε για όλες τις πτυχές της πολιτικής των ενέργειων μεταφορών και όχι μόνο των ενέργειων μεταφορών. Το είπαν ε, και συνάδελφοι Μέσνερ και Κράμερ και ήθελαν να πούν ε, ότι ουσιαστικά αυτά τα θέματα αφορούν ε, όλα τα είδη μεταφορών. Και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύπλοκο το θέμα και από πολιτική και από τεχνική σκοπιά και βάσει αυτού θα πρέπει να δούμε ποια προσέγγιση θα πρέπει να έχουμε εμείς ως Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε ε, με έναν ε, σόφρονα τρόπο, αλλά αποφασιστικά. Δεν θα πρέπει να έχουμε καμία ιδεολογική προσέγγιση, αλλά δεν μπορούμε να παραμείνουμε και στάσιμοι. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε λοιπόν ε, ένα αποτέλεσμα βάση κάποιων στοιχείων αφετηρία θα είναι η κρίση της αγοράς και Φυσικά θα λάβουμε υπόψη και ότι δεν υπάρχουν εδώ κάποια αποκείμενα που μπορούν να χρηματοδοτήσουν άλλους πρωταγωνιστές στο τομέα. Δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε περαιτέρω τη δυσχερή κατάσταση στην οποία λειτουργούν οι αεροπορικές εταιρείες. Δεν ε, είναι τώρα ο καιρός των παχιών αγελάδων για να αφαιρέσουμε αυτές κάποια χρήματα που δεν υπάρχουν. Αυτό το λέω για να διασκεδάσω τις αμφιβολίες, να ξεκαθαρίσω το τοπίο. Είναι δύσκολη η καιρή, αλλά ίσως στο μέλλον είναι ακόμη μεγαλύτερες οι δυσκολίες. Εμείς πιστεύουμε ότι κάποιες δυσκολίες θα μπορούσαν, παραδείγματο χάρη, να προέλθουν από το περιορισμό της χωρητικότητας των αεροδρομίων που θα μπορούσαν να προκύψουν ε, από κάποιες νομοθετικέ διατάξεις που θα περιορίζουν τη χωρητικότητα των διαδρόμων. Παραδείγματο χάρη είχαμε τέτοιες διατάξεις που περιορίζουν την ε, ε, δυνατότητα ε, νυχτερινής προσγείωσης σε ορισμένα αεροδρόμια και αυτό σημαίνει ότι περιορίζεται η χωρητικότητα του αεροδρομίου. Αλλά και εδώ μπαίνω σε ένα έδαφος που είναι πολύ επισφαλές. Μία πιθανή ερμηνεία των ε, υπηρεσιών στο πλαίσιο της ε, γενικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το θέμα των υπηρεσιών. Γιατί εμείς δεν ξεκινάμε από εκεί και αυτό το λέω για να είμαι ξεκάθαρος. Δεν ξεκινάμε από μια πρωτογενή αγορά. Δεν υπάρχει ανάθεση, δεν προβλέπεται ένας διαγωνισμός, δεν προβλέπεται αγοροπολισία ενός αγαθού που δεν είναι δημόσιο. Και θα ήθελα εδώ να κάνω ένα σχόλιο. Τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε τον ορισμό ε, του σλότ της χρονοθυρίδας, οι ανησυχίες είναι πραγματικά τις μερίζονται όλες, γιατί όλα έχουν σημασία, ακόμα και τελείες και τα κόμματα. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε μια δουλειά που να οδεύει προς την κατεύθυνση αυτή. Θα είμαστε πολύ προσεκτικοί, δηλαδή ποτέ δεν αναφέρθηκε ότι οι χρονοθερίδες ε, είναι δημόσια αγωγό, ότι υπάρχει ένας και μόνο ιδιοκτήτης. Λέμε ότι είναι δημόσιας χρήσης αυτό το αγαθό και είναι διαφορετικό γιατί δημόσια ε, χρήση σημαίνει ότι εκεί ομοδοποιούνται τα διάφορα συμφέροντα και ο νομοθέτης που θα κληθεί να εφαρμόσει την ε, νομοθεσία θα πρέπει αυτό να το λάβει υπόψη, να το αξιολογήσει ταυτόχρονα. Όμως ε, έχουμε και άλλη μία κατάσταση. Υπάρχει μία ισορροπία ασταθής αυτή τη στιγμή που δεν θέλει σε ανταγωνισμό τις ε, κανονικές εταιρείες με τις εταιρείες ε, low cost. Οι εταιρείες low cost ε, προτιμούν σήμερα τα περιφερειακά αεροδρόμια, αλλά αν σε κάποια χρόνια η τάση τροποποιηθεί και δηλαδή στραφούν προς ε, τα κεντρικά αεροδρόμια τα οποία σήμερα ε, ουσιαστικά ε, λειτουργούν οι εθνικές εταιρείες, οι εθνικές εταιρείες, εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει με την δευτερογενή αγορά εμπορίας, με τις μεγάλες επενδύσεις που θα μπορούσαν να υπάρξουν εκεί, ποια θα είναι η κατάσταση που θα προκύψει, αλλά εγώ Θέλω να αναφερθώ και σε κάτι ακόμα, στο οποίο αναφέρθηκε και κάποιος συνάδελφος και θα πρέπει να το σκεφτούμε. Η σχέση με την ε, πραγματικότητα, με την εξέλιξη της αγοράς, ε, σε ό,τι αφορά και τις υπόλοιπες υπήρους. Βλέπουμε σήμερα μία εξέλιξη και σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη είναι αρνητική εξέλιξη. Γιατί ενώ πρώτα είχαμε τη Βόρεια Αφρική που ήταν η πρώτη αγορά και ακολουθούσε η Ευρώπη, και τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια και τα βορειοαμερικανικά αεροδρόμια ήταν τα κύρια αεροδρόμια, σήμερα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτές οι δύο περιφέρειες έχουν μείνει πίσω και σε πρώτη θέση βρίσκεται η περιφέρεια της Ασίας και του Ειρηνικού είναι μια περιφερεια που σημειώνεται σημαντική αύξηση και το 2011, με συγχωρείτε, το αεροδρόμιο του Πεκίνου ήταν το δεύτερο σειρά αεροδρόμιο σε φορά τον όγκο των επιθετών μετά την Ατλάντα και ο κατάλογος που έχουμε εμείς για τα αεροδρόμια μας για τα ευρωπαϊκά μας δείχνει ουσιαστικά ότι υπάρχει μια τέτοια μείωση μια τέτοια πτώση. Ένα μόνο ευρωπαϊκό αεροδρόμιο βρίσκεται μεταξύ των πρώτων 25 αεροδρομίων στον κόσμο. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχουν μετακινήσεις ε, και έτσι λοιπόν από αυτή τη σκοπιά πρέπει να γίνουν για κάποιες πολιτικές επιλογές. Εγώ ευχαριστώ όλους όσους πήραν το λόγο. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο τώρα να θίξω όλα τα ζητήματα που θέσατε, αλλά όπως είπε και ο συνάδελφος Φιντάντσα, είναι αλήθεια ότι πρέπει να δράσουμε σε πολλαπλά επίπεδα για να βελτιώσουμε τη χωρητικότητα. Όμως αυτή τη στιγμή έχουμε την δυνατότητα να δράσουμε επί των θεμάτων αυτών. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι θα υλοποιήσουμε νέες δομές, αν τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε ε, για επενδύσεις στο επόμενο δημοσιονομικό τομέα ε, δεν συζητήσουμε θέματα αυτά τώρα, συζητάμε για συνδέσεις στην Ευρώπη και μιλάμε για πόρους. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι οι πόροι θα έρθουν σε ένα, δύο, τρία χρόνια. Όταν κλείσει η περίοδος ε, του δημοσιονομικού προγραμματισμού θα έχουμε μια περίοδο που δεν θα είναι πλέον συμβατή με αυτή την οικονομική προοπτική και απαντούσα έμεσα στον κύριο Σασόλη. Πράγματι, το ε, πεδίο του ορισμού είναι κάπως ολισθηρό, αλλά εμείς ε, όλοι μαζί θα αποφασίσουμε, θα τα σταθμίσουμε όλα τα στοιχεία και θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε και την απόδοση στις διάφορες γλώσσες, θα δούμε και ποιο είναι το νομικό καθεστώς ε, σε κάθε χώρα. Πρέπει να βρούμε σίγουρα μία λύση και θα πρέπει πολύ προσεκτικά να ρυθμίσουμε το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι δεν συμφωνώ με την Επιτροπή στο ότι είναι αρκετά τα δεδομένα ε, των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, γιατί και αυτέ οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές μας δείχνουν που υπάρχουν σύγκρουση συμφερόντων ή που υπάρχει κατάσταση η οποία δεν είναι ολοκληρωτικά διαφανής. Όμως από αυτή τη σκοπιά, συνάδελφος Φώστερ ήδη επανειλημμένος είπε ότι από όσο γνωρίζει Σήμερα δεν πρόκειται για μια αγορά μολυσμένη. Δεν πρόκειται για μια αγορά που αυτή τη στιγμή βλέπουμε κάποιες ε, αρνητικές καταστάσεις που να χρήζουν παρέμβαση. Όμω εγώ νομίζω ότι έχει νόημα να επιζητούμε εμείς τη μέγιστη διαφάνεια. Και να πω και στον κύριο Μπένεν ότι εμείς ε, πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν και οι συνδέσεις με τα περιφερειακά αεροδρόμια, με τις περιφέρειες και από αυτή τη σκοπιά να επιμείνουμε στο δημόσιο χαρακτήρα Δηλαδή, στη δημόσια χρήση των χρονοθερίδων, αυτό επιτρέπει στις εταιρείε να πούν ότι δεν μιλάμε μόνο για αγοροπολισία. Το σλότ δεν είναι μόνο η αγοροπολισία του σλότ που θα καθορίσει το μέλλον των κεντρικών αεροδρομίων και των αεροπορικών συνδέσεων. Τώρα δυσκολεύομαι να αναφερθώ σε όλα τα θέματα που τέθηκαν εδώ. Ζητώ συγγνώμη από όσους ε, τοποθετήθηκαν σε θέματα στα οποία δεν αναφέρθηκα. Όμως εγώ πιστεύω ότι με αυτό το άνοιγμα και με αυτή την ειλικρίνεια με την οποία συνέλεξα τα σχόλια όλων των συναδέλφων, των οποίων σα ευχαριστώ για τη συνεργασία, θα μπορέσω να ε, προσφέρω μια καλή υπηρεσία στο μέλλον των μεταφορών. Ευχαριστώ κύριε Τζες. Τελειώνουμε λοιπόν τη σημερινή μας συνεδρίαση είχε προβληθεί στις 5.30 να ξεκινήσουμε τους συντονιστές. Με συγχωρείτε, ναι, ξαναρχίζω. Η προθεσμία τροπολογιών είναι 12 Σεπτεμβρίου για να ψηφίσουμε στην Επιτροπή τέλος Οκτωβρίου, Οκτωβρίου αρχές Νοεμβρίου και να περάσει την Ολομέλεια την Ολομέλεια το Δεκέμβριο ενδεχομένω. Αύριο θα συναντηθούμε στι 9 και οι συντονιστέ θα συναντηθούν σήμερα το απόγευμα στι 5.30.